Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε τις εργασίες μας. Ε, στην ημερήσια διάταξη έχουμε την ε, ψηφοφορία για μια σειρά εκθέσεων. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να ξεκινήσουμε τις εργασίες του σημερινού πρωινού. Η πρώτη έκθεση που έχουμε να συζητήσουμε. Ε, ένα λεπτό, συγγνώμη, ζήτησε το λόγο ο συνάδελφος Ροϊ, παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, συγχωρέστε με, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ μισό λεπτό την προσοχή σας. Τον επόμενο καιρό και τις εβδομάδες αυτές ε, ήδη συχνά αντιμετωπίζουμε πράξεις κατεξουσιοδότηση που περνάνε από την Επιτροπή και ως, σήμερα αποφασίζουν οι συντονιστές κατά πόσον μπορούμε, θέλουμε ή δεν θέλουμε να τις συζητήσουμε αυτές τις ε, πράξεις. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη διαδικασία, μη δημοκρατική. Θεωρώ ότι και οι βουλευτές, οι μεμονωμένοι βουλευτές, ε, όταν μαζευτούν σε κάποιο αριθμό θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να το θέτουν το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Δεν δέχομαι ένα μικρό περιορισμένος κύκλο να αποφασίζει από μόνο του αν θα πούμε ναι ή όχι. Θέλω να έχω την ε, ευκαιρία να ψηφίζω. Δεν είμαι δευτέρα κατηγορία, ούτε τρίτη κατηγορία βουλευτή. Δεν το δέχομαι. Γι' αυτό κυρία Πρόεδρε σα ε, παρακαλώ να ψηφίζουμε στι επόμενε συνεδριάσει ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Γιατί αυτό αφορά όλη την Επιτροπή. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε και σας παρακαλώ να βρούμε μία διαδικασία, όχι εντάξει να το ζητάει ένας μόνος βουλευτής από μόνος του, όχι, αλλά ένας συγκεκριμένος αριθμός βουλευτών να έχει το δικαίωμα να θέσει ένα τέτοιο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σας παρακαλώ να το ψηφίσουμε αυτό σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις. Όχι σήμερα, πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία. Αλλά αν μας αφαιρείτε το δικαίωμα αυτό, πρέπει πραγματικά να ζητήσουν να το ψηφίσουμε. Σα παρακαλώ να το κάνουμε σε μία από τι επόμενε συνεδριάσεις, να το θέσουμε στην ημερήσια διάταξη, να έχουμε την ευκαιρία να προετοιμαστούμε. Είμαι πάρα πολύ αγανακτισμένος. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτά τα παιχνίδια είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία τελικά μα εκθέτουν και στο εκλογικό μα κοινό, να σα το πω και έτσι. Τουλάχιστον να έχουμε την ευκαιρία να το ψηφίσουμε. Τουλάχιστον αυτό. Μπορεί τελικά η ψηφοφορία να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που επιθυμώ εγώ, αλλά το να ψηφίσω είναι ένα δικαίωμα που δεν μπορεί να μου τα αφαιρέσει κανένα. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Ντοέλ. Έχει ζητήσει το λόγο ο συνάδελφο Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Καταλαβαίνω αυτά που λέει ο συνάδελφο κύριε Ρόιλ. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας υποδείξω το εξής. Οι συντονιστές εκλέγονται από τα μέλη της ομάδας τους. Εκπροσωπούν δε την ομάδα στις συνεδριάσεις των συντονιστών. Άρα δεν είναι θέμα ότι κάποια τυχαία άτομα παίρνουν αποφάσεις. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, όπως είμαι βεβαίως ότι θα πείτε και εσείς κυρία Πρόεδρε προς τον κύριο Ρόιλ, ε, που θα μας οδηγήσει σε μια συμφωνία για τη διαδικασία για τις πράξεις εξουσιοδότηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, μάλιστα. Και στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο εν γέννη θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των ε, πράξεων που λαμβάνουν χώρα μέσω επιτροπολογίας. Και αυτό φυσικά ε, προαπαιτεί και κάποιο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αλλά να υποδείξω και στον συνάδελφο ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι μέσα στις ομάδες με τους οποίους μπορούν να δράσουν οι βουλευτές από κοινού ή και μεμονωμένα, για παράδειγμα η συλλογή 40 υπογραφών, για να θέσουν τέτοια θέματα, να διαβεβαιώσω δε και τον κύριο Ρόιλ ότι με απασχολεί και όλο ο ιδιαίτερος το θέμα αυτό και εμένα. Ευχαριστούμε για να απαντήσω στον συνάδελφο που παρενέβηκε μετά θα περάσουμε στην ψηφοφορία εντός της Επιτροπής. Η ΤΡΕ με τη γενική διαδικασία που θα υιοθετήσουμε για τις κατεξουδότηση πράξεις. Θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε και λίγο την λήψη απόφασης. Φυσικά ο κάθε συντονιστής θα αναφέρει στην δική του ομάδα τις εργασίες μας σε αυτή τη μεταβατική περίοδο και ενώ αναμένουμε να επιτευχθεί μια κοινή στάση για το πώς θα προσεγγίσουμε το θέμα των κατεξιδότηση πράξεων, οι συντονιστές αποφασίζουν φυσικά βάσει των πλειοψηφίων των ομάδων στις οποίες ανήκουν ε, και βάσει των οποίων ο ε, θα τεθεί ξανά το ερώτημα στην Ολομέλεια. Ε, ευχαριστούμε τον συνάδελφο Ρόλη για την παρεμβασή του και τον συνάδελφο Τσίτσεστερ. Περνάμε λοιπόν ε, στην πρώτη έκθεση. Ο συνάδελφος Ρόιλ, συγγνώμη. Να ξέρω μόνο θέλω, γιατί αυτό το θέμα θα μπει σαν θέμα σε συνεδρίαση της ομάδας, της Επιτροπής. Θέλω να μπει στην ημερήσια διάταξη στην ημερήσια διάταξη. Εγώ νομίζω ότι ζητάτε κατά πόσο θα συμπεριλάβουμε το θέμα αυτό της τάση μα για τις κατεξοδότητες πράξη στην ε, ημερήσια διάταξη. Ναι, μπορούμε. Ευχαριστώ, συνάδελφε Ραπόρτο. Περνάμε στην έκθεση ΡΕΜΕΚ. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Ρέγω. Να επαληθεύσουμε πρώτα τη χρήση της, των καρτών ψηφοφορίας. Ε, είστε όλοι έτοιμοι να ψηφίσετε, παρακαλώ. Ωραία, κλείνει η ψηφοφορία. Έχουμε 30. 30 παρόντες αυτή τη στιγμή. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 15 και 16 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 28 τροπολογία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ το δεύτερο τμήμα δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε λοιπόν τροπολογία 29 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία να ελέγξουμε την 29 πολύ ωραία Πρώτο τμήμα ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Κλείνει η ψηφοφορία. 5 υπέρ 35 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60 το δεύτερο τμήμα του τροπολογίας 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κάποια σύγχυση έχει δημιουργηθεί. Τροπολογία 8. Λοιπόν, του έλκυνη σελίδα 5. Βρισκόμαστε στην τροπολογία 8 της Επιτροπής Προπολογισμού. Τροπολογία 8 της budget για το ΕΛΚ σελίδα 5. Σελίδα 5, τροπολογία 8. Τη βρήκατε? Ωραία. Είμαστε στο σημείο. Λοιπόν, τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται φαίνεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 8. Τροπολογία 8 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54-55 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά 56 καταπίπτει γιατί εγκρίναμε την 10 Συνεπώς η 56 καταπίπτει και περνάμε στην 58. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 3. Πέραση ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 37 και τροπολογία 6 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 38, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 39 ή 40 συγγνώμη 40 ζητώ συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία για το σύνολο άρχεται η ψηφοφορία διαδικαστικό Θα ήθελα να ελέγξουμε την ψηφοφορία για την τροπολογία 3. Την τροπολογία 3. Γιατί θεωρώ ότι προκλήθηκε μία σύγχυση. Σας παρακαλώ να επανέλθουμε στην ε, τροπολογία 3 και να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. rejeté. On a voté au... Scusi relatore, l'emendamento 3 su cosa? Sul budget? Την τροπολογία 3, ποια ε, budget? 3 budget ή... Ναι, είναι δική... είναι δική μου τροπολογία για το 8 άρθρο 2 παράγραφος 1 για τον προϋπολογισμό. Τροπολογία 3 του συγγητή. Ζητώ συγγνώμη, ο κύριος εισηγητής ε, είχε απορριφθεί η τροπολογία 3. Είχε απορριφθεί. άρθρο 2 παραγραφός 1 τροπολογία 3 απορρίφθηκε όπως καταλαβαίνετε εκτός από το ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε τους κανόνες ψηφοφορίες αυτό θα επηρεάσει και τις επόμενες ψηφοφορίες διότι ανάλογα με αυτό επειδή καταπίπτει ψηφίσαμε και άλλα σημεία στη συνέχεια. Το 7, το 43, συνεπώς δεν μπορούμε να επανέλθουμε στην ψηφοφορία, ζητάμε συγγνώμη, μπορούμε να το αλλάξουμε στην Ολομέλεια. Τελική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Για το ψήφισμα αυτό έχουμε 38 υπέρ, 4 κατά, 5 αποχές. Για την έκθεση, συγγνώμη, και τώρα ψηφι... Ε, ψηφίζουμε για το ψήφισμα, άρχεται ψηφοφορία. Ωραία, λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας, 37 υπέρ, 5 κατά και τελική ψηφοφορία, τελευταία ψηφοφορία, Πέρα ψηφοφορίας. Ραπόρτο Τόια. Έκθεση Τόια. Συμβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τοπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τοπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τοπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 26. Πέρας της ψηφοφορίας. «25 υπέρ, 21 κατά δεκτή, 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34, 33 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 34. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την τροπολογία 34. Emendamento eh, chiuso, approvato ampiamente, grazie. Emendamento 35, a favore, contrari, astenuti, approvato. Compromesso 7, a favore. Συμβιβαστική 7, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 39, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 68 παρακαλώ. 25 υπέρ 18 κατά δεκτή. Η 70 τώρα υπέρ κατά. Αποχές δεκτή. 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 90 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 90 παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. 36 κατά 7 υπέρ, 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 99 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, α, Κοιτάξτε θα ξαναψηφίσουμε, δημιουργήθηκε μια παρανόηση για την 100. Ποιοι είναι υπέρ της 100. Κατά αποχές δεκτή. 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 104 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 110 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 112 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 113 υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 118 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 119 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 120 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 123 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ψηφίζουμε τελική ψήφος πλέον. Πέρας της ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 4 κατά, 4 αποχές, συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας, έχετε το λόγο. Ε, να ευχαριστήσω και εγώ, λέει η κυρία Τόια, με τη σειρά μου στους συναδέλφους, γιατί η έκθεση, έτσι όπως είναι τώρα σε σχέση με το πώς ξεκίνησε, είναι άλλο πράγμα. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν και ευχαριστώ και τους συνεργάτες μας, ε, βοηθούς, ε, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κυρία Τόρια. Τώρα πηγαίνουμε στην ε, γνωμοδότηση του κυρίου Ράνστορφ. Περνάμε στην τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές Αρχιτελεκτρονική ηλεκτρονική ψηφοφορία. για την 8 Παέρας ψηφοφορίας 19 υπέρ 19 υπέρ, 18 κατά, 6 αποχές. Πολύ ωραία εγκρίνεται η τροπολογία 8. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ να ελέγξουμε τη 15 παρακαλώ άρχιτε ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 22-22. Απορρίπτεται. Η 15, έτσι, όχι 14 όπως είπε ο Πρόεδρος. Ε, είμαστε στην 16, περνάμε υπέρ. Κάτα, αποχές, φαίνεται να απορρίπτεται, αλλά δεδομένου του προηγούμενου αποτελέσματος προτείνω να ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία για την 16. 16. Τροπολογία 16. Αυτήν ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας 19 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 21 ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας 22 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται ή 21. 22 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 26. Να ελέγξουμε την 24. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία 19 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, ωραία λοιπόν 42 υπέρ, 2 κατά, συγχαρητήρια στον συνάδελφο κύριο Ράνστορφ. Τελείωσε η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ να περιμένουμε πέντε λεπτά ώστε να φύγουν από την αίθουσα όσοι θέλουν να φύγουν και θα συνεχίσουμε με την έκθεση Rubik. Όποιος είναι να φύγει παρακαλώ να το πράξει ταχαίως.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 Passiamo piano di azione Πρόγραμμα δράσης λοιπόν, επιχείρηση του 2020. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Ρουμπίχ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ένα θέμα όπου ουσιαστικά στην Ευρώπη ανησυχούμε ιδιαίτερως η ανεργία των νέων. Δραματικά επίπεδα έχει φτάσει και γι' αυτό λοιπόν όταν υπάρχουν τόσο πολλοί άνεργοι και δεν υπάρχουν εργοδότες, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να τους ε, εκπαιδεύσουμε, πώς μπορούμε να ε, προωθήσουμε την ανεξαρτησία τους και πώς μπορούμε την καταστροφή αυτή της τεράστιας αυτής ανεργίας να την καταπολεμήσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ιδιαίτερως οι νέοι, οι νέοι επιχειρηματίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ε, καταδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δημιουργούν θέσεις εργασίας. Τέσσερα εκατομμύρια ανά έτος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι η επιχειρηματίες. Οι επιχειρήσεις που ε, είναι, έχουν ε, διάρκεια ζωής μικρότερη των πεντε ετών δημιουργούν ιδιαίτερα πολλές θέσεις απασχόλησης. Από την άλλη, αποθαρρύνεται ο κόσμος από το να αναπτύξει επιχειρηματική δράση. Και τα τελευταία τρία χρόνια βλέπουμε ότι το ποσοστό των νέων επιχειρηματιών έχει πέσει από 45% σε 37%. Υπάρχει λοιπόν μια αποθάρρυνση από την επιχειρηματικότητα, από την πρόσληψη νέων ανθρώπων και όλα αυτά φυσικά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Στην τελική ανάλυση μπορούμε να πούμε βέβαια ότι 37% των πολιτών παρόλα αυτά ε, θέλουν να είναι αφεντικά του εαυτού τους, αν θέλετε. Αναλαμβάνουν τους κινδύνους που συνεπάγεται μια νέα επιχείρηση. Άρα έχουμε 20.000 ε, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Αν προωθούσαμε λοιπόν αυτές τις επιχειρήσεις δεν είχαμε προβλήματα με την ανεργία. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να προωθήσουμε τα άτομα αυτά που θέλουν να είναι ανεξάρτητα προκειμένου να δείξουν το θάρρος που χρειάζεται και να προσλάβουν κάποιον είναι κεντρικό το ερώτημα του ποια είναι τα κίνητρα τα οποία θα πρέπει να δώσουμε στα εκατομμύρια επιχειρηματίες που θα μπορούσαν ενδεχομένω κάποιον να προσλάβουν, κάποιον να απασχολήσουν. Αντιθέτως λοιπόν με τις άλλες εκθέσεις που έχουμε καταρτήσει σε ό,τι αφορά τις μικρομεσίες επιχειρήσεις, στη δική μου έκθεση θέσουμε το επίκεντρο στην ε, επιμόρφωση, στην κατάρτιση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική κατάρτιση. Υπάρχουν σε κάποιες χώρες ε, κάποια πιλωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα όπου στο σχολείο διδάσκεται ακόμα πώς ε, μπορεί κανείς να διοικεί μία εταιρεία. Θυμάμαι και στον υπηαγωγείο που είχαμε για παράδειγμα ένα μαγαζί πλαστικό που έπαιζε κανείς στον έμπορο, πώς ε, πουλάει, πώς αγοράζει ε, γάλα, γιαούρτια. Τι να σας πω, ήταν πάρα πολύ δημοφιλές αυτό το παιχνίδι, ίσως γι' αυτό τελικά και εγώ να είμαι ε, εξελίχθηκα σαν εξάρτητο επαγγελματία, αλλά αυτό που είναι γεγονός είναι ότι αυτά τα έργα τα οποία συνδέονται με επιχειρήσει με πανεπιστήμια, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Υπάρχουν πάρα, πολλές, ε, πολλά πανεπιστήμια, όπου για παράδειγμα υπάρχει αυτόνομη διαχείριση τη βιβλιοθήκη, για παράδειγμα, για να δείξει ακριβώ στους φοιτητές ότι υπάρχει κάποιο νόημα στην αυτόνομη διαχείριση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα μέχρι το 2015 τα κρατημέλη μας να υποχρεωθούν να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ε, συμπερίληψη της επιχειρηματικής κατάρτισης στο σχολικό πρόγραμμα και στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι το πιο βασικό θέμα το οποίο ζητούμε. Να διαμορφώσουμε με καλύτερο τρόπο την εκπαίδευση τους στα σχολεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους ε, απασχολούμενους. Να υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι να γνωρίζουν τι συνεπάγεται η εργοδοσία, τι υποχρεώσει, τα δικαιώματα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Η πρόκληση τη εκπαίδευση, στο δεύτερο σημείο. Χτε συνεχάρη τον ε, ε, Επίτροπο Τατζάνη, γιατί το πρόγραμμα Εράσμους για τους νέους επιχειρηματίες έχει σημειώσει τεράστια ε, επιτυχία σε χώρες με μεγάλη ανεργία. Πολλοί νέοι έχουν δεχτεί αυτή την πρόκληση του να πάνε σε μια άλλη χώρα, σε ένα άλλο κράτος μέλος και εκεί να κάνουν μια πρακτική σε μια άλλη επιχείρηση, να δουν πώς την πράξη λειτουργεί μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι πάρα πολύ καλό πρόγραμμα αυτό και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να θέσουμε το στόχο των 10.000 συμμετεχόντων ανά έτος. Είναι μεγάλη η επίτραση ενός τέτοιου προγράμματος και νομίζω ότι αυτό θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην Ευρώπη προκειμένου να υπάρξει η κατάρτιση των νέων και να επιστρέψουν μετά οι νέοι με νέα προσόντα στην χώρα τους. Χρειαζόμαστε ασφαλώς και κονδύλια. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να θέσει νέα επίκεντρα πολύ καλό και το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Νομίζω ότι και αυτό θα μπορούσε μαζικά, δραματικά να συμβάλλει εδώ στην προώθηση αυτού του νεαρού επιχειρηματικού πνεύματος. Εδώ στην Αστρία με τα συνδικάτα έχουμε χρησιμοποιήσει και εφαρμόσει πάρα πολύ καλά αυτά τα κίνητρα και βλέπουν τα συνδικάτα ότι σε συνδυασμό με την εργοδοσία σημειώνονται πάρα πολύ καλά αποτελέσματα με τους μετανάστες, με τους νέους ε, εργαζομένους. Και εδώ το Εράσμος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι τεράστιο το δυναμικό εδώ. Και φυσικά στο EIT νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να προωθηθεί και η επιχειρηματική κουλτούρα σε ό,τι αφορά τους νέους επιχειρηματίες. Το θέμα είναι η αξιοποίηση το, της γνώσης που προκύπτει από τα ερευνητικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό προωθεί και η Επιτροπός Βασιλείου, αλλά η τεχνολογία της εκμάθησης, της διδασκαλίας εδώ στην Ευρώπη είναι παροχημένη. 25 χρόνια είναι παλιά, αν θέλετε, πριν από 25 ετία ήταν. Ακολουθούμε τι ίδιε διδακτικέ ε, πρακτικέ στα πανεπιστήμια όπω και πριν από 25 χρόνια. Θα πρέπει αυτά να προωθήσουμε από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, από κοινού με την Επιτροπή Βιομηχανία, προκειμένου στον τομέα αυτό να δώσουμε μια ισχυρή όθηση. Αλλά νομίζω ότι στη τελική ανάλυση θα πρέπει να κοιτάξουμε το σχέδιο δράσης ε, για τους επιχειρηματίες και το Small Business Act. Να το δούμε με νέο μάτι. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία μπορεί να συμβάλλει παραπάνω προς την κατεύθυνση αυτή. Το θέμα είναι να μετρήσουμε πόσο χρόνο χρειάζεται σήμερα η δημιουργία μιας επιχείρησης, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί ο χρόνος έγκρισης ε, μιας επιχείρησης και το One Stop Shop είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια ενιαία θηρίδα μέσω της οποίας μπορεί να γίνουν όλα τα βήματα. Και φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η δημιουργία και η μεταφορά επιχειρήσεων γιατί σε οικογενειακές επιχειρήσεις ε, είναι πολύ συχνά βλέπουν πόσο δύσκολο είναι να τρέξει μια επιχειρήση και προτιμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλο τομέα. Γιατί πολύ απλά, και κλείνουν οι εταιρείε γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει διάδοχος. Ιδιαίτερα σε περίπτωση που υπάρχει και καδημαϊκή μόρφωση, πολλοί θεωρούν ότι δεν αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί η επιχείρηση των γονέων και έτσι χάνονται θέσει εργασία. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Η δεύτερη εταιρεία επίσης, η δεύτερη ευκαιρία για παλιές εταιρείες οι οποίες κλείνουν γιατί δεν έχουν για παράδειγμα άλλο αντικείμενο. Ε, παλαιοί όμιλοι οι οποίοι διαλύονται και επιχειρήσεις οι οποίες ε, αναγκάζονται να συνεχίζουν να πληρώνουν τους ε, οδότες τους τους εργαζομένους τους γιατί δεν μπορούν να τους απολύσουν, δεν μπορούν να πάρουν ε, πιστώσεις και τελικά φυσικά πτωχεύει η εταιρεία και τελικά παρόλα αυτά καταλήγουν στον δρόμο οι εργαζόμενοι. Άρα τέτοιες εταιρείε πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τις προστατεύσουμε και αυτές και τους εργαζόμενους σε αυτές για σε τελική ανάλυση και εδώ θα κλείσω. Το θέμα είναι το εξής. Χρειαζόμαστε υποδείγματα, παραδείγματα Έχουμε παραδείγματα, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον δυναμικό των γυναικών. Οι γυναίκες, νομίζω, χρειάζονται πάρα πολύ ελευθερία στην κατανομή του χρόνου, στην αυτοδιάθεσή τους. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, γιατί μόνο το 34% των ε, αυτοαπασχολούμενων στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια ξεσορρόπηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν σχετικά προγράμματα. και οι γυναίκες επιχειρηματίες χρειάζονται μεγαλύτερη ελευθερία. Θα πρέπει τα εμπόδια που υπάρχουν για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας και σε ό,τι αφορά αυτή την αυτοδιάθεση, την ανεξαρτησία τους, να καταργηθούν. Ίσως μια μέρα, να καθαριθεί μια ημέρα ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας. Ίσως την 1η Μαΐου, ίσως αυτό θα ήταν ένα καλό παράδειγμα για την κοινωνική εταιρική σχέση. Ότι μόνο από κοινού οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μπορούν να είναι δυνατοί για να καταπολεμήσουν τα εμπόδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ίσως και 30 Απριλίου δεν έχω εγώ ένσταση. Σημαντικό είναι να μην θέσουμε στο επίκεντρο τις διαφορές, τα σημεία, τα ακαθόδη, αλλά τους κοινούς τους στόχους. Προς αναζήτηση φυσικά κοινών στρατογικών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στην Ευρώπη να βρούμε κοινούς στόχους. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό για την επόμενη γενιά να δημιουργήσουμε ένα κλίμα αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης. Ότι στην Ευρώπη μπορεί κανείς να είναι αυτόνομος να απασχολείται σε μια οικογενειακή επιχείρηση και να στεφτεί με επιτυχία επαγγελματικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτός μικροφώνου μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο εισηγητή για τη συμβολή του, για τις προτάσεις του. Αυτή η ημερίδα μου φαίνεται εξαιρετική ιδέα. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα η οποία πλήττεται σκληρά από την κρίση. Υποφέρει από ανεργία, από τον όλο πληθυσμό. Χρειάζεται ωστόσο να γίνει πιο ανταγωνιστική, να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. Φυσικά η κατάσταση διαφέρει σε συνάρτηση με τη χώρα. Αυτά τα κριτήρια λοιπόν εξυγχρονισμού των πρακτικών και της κοινή χρήση των λύσεων είναι λίγο παλιές όπως φαίνεται ανάλογα με την κατάσταση του κάθε κράτους μέλους. Η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού σχεδίου μπορεί να αποτελέσει λύση πράγματι. Η μείωση του χρόνου και των χρόνου που χρειάζονται για τη δημιουργία μιας ε, επιχείρησης φυσικά είναι εμπόδια στη δημιουργία επιχειρήσεων και στην επιχειρηματικότητα ορισμένες επιχειρήσεις ε, καταφεύγουν στις ε, εξαγωγές και κάθε άδεια παίρνει πολύ χρόνο. πρόβλημα από οικονομικής άποψη είναι η ανεπάρκεια των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις. Είναι κρίσιμη σημασία. Χθες πάλι στην Επιτροπή Ήτρε είπαμε ότι για μια ισπανική επιχείρηση τα επιτόκια είναι διπλάσια από ό,τι στη Γερμανία. Οι επιχειρήσεις δηλαδή καταβάλουν πολύ περισσότερο κόστος δανεισμού. Και όσον αφορά την ανεργία των νέων στην Ισπανία, πολύ συχνά οι νέοι έχουν εξαιρετική εκπαίδευση, είναι μεταξύ 25 και 30 χρονών και χρειάζονται βοήθεια. Χρειάζονται πρόσβαση σε πίστοση Αυτή η νέοι ανεργή. Πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα ώστε να μην μένουν ευάλωτοι χωρίς καμία προστασία ε, ενώπιον των πιστώσεων. Μιλήσαμε για το Εράσμους. Εγώ πιστεύω ότι το Εράσμους βοήθησε στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών, βοήθησε στην ε, ανάπτυξη στην Ευρώπη, αποτέλεσε σημαντική κινητήριο δύναμη για τον εξευρωπαϊσμό. Ε, το μείωση λοιπόν αυτών των κονδυλίων είναι απαράδεκτη. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μια υπεράθρωπη προσπάθεια για να πούμε σαφώς στο Κομισιόν και στο Συμβούλιο ότι η αυτοαπασχόληση μπορεί να αποτελέσει λύση για την κρίση αλλά θα χρειαστούν τα κατάλληλα μέσα. Θα χρειαστεί να αγωνιστούμε και κυρίως να αποφύγουμε οποιαδήποτε διαστρέβλωση και διαφορά μεταξύ χωρών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματο του κυρίου Κρόιτσμαν, ο οποίο είναι σκιώτης εισηγητής τη ομάδα των φιλελευθέρων, ο οποίο δυστυχώ ε, βρίσκεται σε μια άλλη επιτροπή και ψηφίζει. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω το σχέδιο έκθεσης ε, ψηφίσματος ε, του κυρίου Ρούμπιχ που περιλαμβάνει πολλές καλές ιδέες σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και ε, να πούμε ότι η οικονομική κρίση αποθαρρύνει πάρα πολλούς Ευρωπαίους από το να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση και οι πιο πολλοί τομείς πολιτικής που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά σίγουρα θα πρέπει να εντοπίσουμε με συντονισμένο τρόπο τις βέλτιστες πρακτικές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, ε, ο τομέας της ε, εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν στην εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που θα πρέπει να διδαχτούν στο σχολικό πρόγραμμα. Ω τώρα είναι σχεδόν απολύτω απόντα τέτοια στοιχεία. Τα σχολεία όπου κάνουν τα σχολεία συγκεκριμένες προσπάθειες, αυτό αποδίδει καρπούς. Αυξάνεται το ποσοστό 3 έως πέντε φορές παραπάνω των ε, μαθητών που ε, ιδρύουν αργότερα επιχειρήσεις. Ε, επίσης θα ήταν θεμητό να δημιουργηθούν ε, θέσεις ε, πρακτικής ε, σε πραγματικές επιχειρήσεις στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Κατά δεύτερον, υποστήριξη έναρξης νέων επιχειρήσεων. Υποστηρίζουμε φυσικά όλα τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνούμε όμως με τον εισηγητή ότι οι περικοπές του προγράμματος COSME κατά 14% είναι απαράδεκτες. Η μείωση επίσης του γραφειοκρατικού άχθους είναι πολύ σημαντικός ε, παράγοντας για την πρόθεση των επιχειρήσεων. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν εκπληρώσει τις παλαιότερες δεσμεύσεις για τη μείωση όλου του γραφειοκρατικού άχθους που συνεπάγεται η έναρξη μιας επιχείρησης. Χρειαζόμαστε λοιπόν φιλόδοξα φιλόδοξου στόχους στο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Ρόντε. Ε, το λόγο έχει η συνάδελφο κυρία Φόρντ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω αρχικά ότι είναι εξαιρετικό που αυτή η Επιτροπή αυτού του Κοινοβουλίου επιτέλους εστιάζεται στην επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρηματίες είναι το κλειδί της επιτυχούς ανάπτυξης της δημιουργίας επιχειρήσεων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας εξορισμού. Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν όταν βρίσκουν νέες ευκαιρίες και ε, είναι επιτυχής ως επιχειρήσεις. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες μας να λειτουργούν σε έναν παγκόσμιο ανταγωνιστικό κόσμο Τώρα όσον αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, πιστεύω ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να εστιαστούμε και επιμένω εδώ και τέσσερα χρόνια σε αυτό το κοινοβόλιο για το πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο. Ε, υπάρχει αυτή η λίστα με τους δέκα πιο επαχθείς ε, ευρωπαϊκούς νόμους και θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι αυτές που πρέπει να εξαιρέσουμε το ταχύτερο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ρύθμιση, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία από τις μικρές προς τις μεσαίες και μετά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Θα πρέπει ωστόσο να προσέξουμε τα ζητήματα που εξετάζουμε σε θέματα αρμοδιότητων. Ναι, μπορούμε να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές, η κατάρτιση είναι σημαντική συχνά βλέπω ότι η κατάρτιση και η υποστήριξη της επόμενης γενιάς, η επανεκπαίδευση σε νέες δεξιότητες ε, παρέχεται καλύτερα σε τοπικό, σε εθνικό επίπεδο, γιατί πρέπει να είναι κανείς βέβαιος ότι παρέχει τις δεξιότητες, τις ικανότητες για τις δουλειές που υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Συχνά λοιπόν βλέπω προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαρθρωτικά κονδύλια ή την ε, χρήση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και παρατηρώ ότι δεν φέρνουν τα αποτελέσματα που θα έπρεπε, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε σχέση με το αν τα χρήματα είχαν διοχετευτεί μέσω ενός τοπικού προγράμματος, ενός εθνικού προγράμματος, ώστε να διοχετευτούν καλύτερα σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τι ε, βέλτιστε πρακτικέ και όσον αφορά το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, μερικέ φορέ ε, αυτό διευκολύνει τι λιγότερο ανταγωνιστικέ εταιρείε να ε, μετακινούν θέσει εργασία. Το σχόλιο σα το να δώσουμε νέα κίνητρα για επιχειρηματική φιλοσοφία. Κατά την άποψή μου, υπάρχουν ήδη πολλά κίνητρα χρειαζόμαστε ε, και ένα νέο οργανισμό, αλλά η επιχειρηματικότητα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε οποιοδήποτε κίνητρο. Το κίνητρο είναι να δώσουμε γνώση στις νέες αγορές, στις νέες επιχειρήσεις. Όχι απλά κίνητρο δηλαδή για τις επιχειρήσεις, κίνητρο για τα πάντα. Ωραίες είναι οι όμορφες διατυπώσεις, τα όμορφα λόγια, αλλά στη δικό μου κράτος πρόσφατα τα δάνεια, οι χορηγήσεις, τα δάνεια που δόθηκαν για startup εταιρείε ε, δόθηκαν σε γυναίκες. Αλλά οι γυναίκες ήδη είναι εξαιρετικές επιχειρηματίες. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω βοήθεια. Πολλές φορές ηγούμαστε επειδή τολμάμε τις προκλήσεις ε, με διαφορετικό τρόπο. Όσον αφορά το κόσμο, Υπάρχουν και ανησυχίε για το κόσμο, αλλά γενικά θέλουμε ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάζεται στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Και αντί για αυτό, έχουμε ένα πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που ενσωματώνει την κοινή γεωργική πολιτική σε να πηγαίνει πίσω. Ενώ θα έπρεπε να εστιαζόμαστε στο μέλλον και στο πώ θα βοηθήσουμε του επιχειρηματίε μα. Θα ήθελα λοιπόν να γίνεται αναφορά αυτού. Με τα εγγύηση για τους νέους με ανησυχεί δεν θα λύσει τα προβλήματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ακούγεται ωραία, αλλά το να εκπαιδεύει κανεί ανθρώπου για εργασίε που πρόκειται να εμφανιστούν είναι κάτι που γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο τη εγγύηση για του νέου. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η συνάδελφο Χιμπνερ. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η επιχειρηματικότητα μετά την ενέργεια και την ψηφιακή ατζέντα θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας και να σας πω ότι εγώ έχω αντιμετωπίσει προβλήματα σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, ακόμα και στην ίδια μου την οικογένεια. Προσπαθούν τα παιδιά μου να γίνουν επιχειρηματίε. και ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η ενεργεία μεταξύ των νέων είναι πάρα πολύ ψηλή. Όχι όμω επειδή δεν υπάρχει διάθεση δημιουργικότητα και ανατομίας. Είναι πάρα πολύ δημιουργική η νέα γενιά, αλλά υπάρχουν εμπόδια. Υπάρχουν εμπόδια. Δεν είναι εύκολη πρόσβαση στα ε, στις πιστώσεις και επίσης υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία. Να θυμόμαστε ότι αυτά που δημιουργούνται τώρα ουσιαστικά διαρκούν 2-3-10 χρόνια. Ε, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει νομική βεβαιότητα και η κατάσταση να αλλάζει κάθε 2-3 χρόνια. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Αμερική. Κατά μέσο όρο οι νέοι αλλάζουν καριέρα ε, κάθε μάλλον δύο-τρει φορέ στην ζωή του. Ενώ στην Ευρώπη υπάρχει αντίληψη ότι πρέπει κανεί να μένει στην ίδια θέση μια ολόκληρη ζωή. Θα πρέπει ίσω να δείξουμε στον κόσμο ότι ιδιαίτερα σε δύσκολε εποχέ ε, κρίση πρέπει κανεί να διακινδυνεύει και να παίρνει ρίσκα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα κάνει κάτι εντελώ διαφορετικό, κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας ε, του ατόμου. Ένα πρόγραμμα λοιπόν το οποίο θα έδινε μια νέα διάσταση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, σε έναν τελείως, εντελώς καινούριο τομέα, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να υποστηρίξουμε. Ξέρουμε όλοι ότι ε, πολύ σύντομα θα έχουμε έλλειψη 2 ε, εκατομμυρίων ε, ειδικών στον τομέα του IT στην Ευρώπη. Ίσως θα πρέπει να το υποδείξουμε αυτό στους νέους, ότι κοιτάξτε, αυτό είναι ένας τομέας ο οποίος θα αντιμετωπίσει έλλειψη στο μέλλον. Δεν είναι μόνο ε, η πολιτική. Δεν είναι μόνο η ψυχολογία, για παράδειγμα, τομείς ε, όπου χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Όχι, τεχνική τομείς. Αυτό έχει να κάνει και με την ψηφιακή ατζέντα, με τον κυβερνοχώρο που αναπτύσσεται ταχύτατα. Αυτό λοιπόν να το υποδείξουμε στους νέους είναι το μέλλον πραγματικά. Ας επικεντρωθούμε επίσης και στην σταθερότητα των νομικών ε, κανονισμών και στην χρηματοδότηση των νέων επιχειρήσεων με χαμηλά επιτόκια. Και ναι, η εκ νέου κατάρτιση για να αλλάξει κανείς εντελώς κλάδο στην επιχειρηματικότητά του. Ευχαριστώ πολύ. Το συνάδελφο έχει... Ο λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Πρόντι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο κ. Ρούμπιχ ε, για τη σύνταξη αυτού του εγγράφου που είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ με το όσα είπε. Δεδομένης και της συζήτηση που κάναμε λεπτομερώς και χθες ε, για τις διάφορες πτυχές της επιχειρηματικότητας ε, θυμάμαι που συζητήσαμε για την επανεκβιομηχάνηση του Νότου της Ευρώπης. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, καθώς και η συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη. Εκεί Είδαμε το τεράστιο φάσμα προβλημάτων αλλά και δυνατοτήτων που υπάρχουν για τους επιχειρηματίες. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω μόνο ένα πράγμα στα όσα υπόθηκαν με τα οποία συμφωνώ. Θεωρώ ότι ειδικότερα για τους νέους είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα ότι σημασία δεν έχει μόνο η σύσταση μιας επιχείρησης που μπορεί να λειτουργήσει σωστά αλλά και της προσφοράς μιας επιχείρησης στην κοινότητα. Με αποτέλεσμα η κοινότητα να αναγνωρίζει αυτή την επιχείρηση ως κοινό αγαθό. Πιστεύω λοιπόν ότι η προσπάθειά μας πρέπει να εστιαστεί στο να επιδιώξουμε, να δώσουμε και αυτή την πτυχή να την καταλάβει ο κόσμος γιατί έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές διάφορα σκεπτόμενοι ότι η μεταποιητική βιομηχανία είναι κάτι ξεπερασμένο και ότι συνεπώς δεν αξίζει ενδεχομένως να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό το τομέα της βιομηχανίας γιατί ούτως ή μπορούμε να τη στείλουμε σε άλλες χώρες και οδηγηθήκαμε στην καταστροφή της βιομηχανίας μας. Εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε αυτή τη συζήτηση και να προσφέρουμε στους νέους μια άλλη εικόνα ότι μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί με γνώμονα την κατάρτιση, την απασχόληση που προσφέρει, την ευημερία που δημιουργεί και βάσει μιας τέτοιας προσδοκίας ε, η κοινωνία ενδεχομένως θα αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα. Να γίνει και μια πρόταση οργάνωσης ε, που, διαφόρων αξιών που μπορεί να είναι και πιο σημαντικές από τα κέρδη ως αξία. Δηλαδή αναφέρομαι εδώ στην κοινωνική ευθύνη μια επιχείρηση, αλλά και σε κάτι ακόμη πιο ευρύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συναδέλφο κύριο Πρόντι. Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Τρότμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι έρχεται σε πολύ κατάλληλη στιγμή αυτή η έκθεση και θα ήθελα να μοιραστώ με τους συναδέλφους κάποια πράγματα που με προβληματίζουν όπως τα έμαθα πρακτικά σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης και ειδικότερα όσον αφορά τη δημιουργία ή την ανάκαμψη των δραστηριοτήτων. Πρώτη διαπίστωση. Ενίοτε έχουμε σκεφτεί ότι η δυνατότητα της αυτοαπασχόλησης είναι λύση για την ανεργία. Συνέβη στη χώρα μου, οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις επιτυχίας είναι κατάρτιση, ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο, το οποίο πρέπει να έχει επαληθευτεί πριν ζητήσει κανείς πίστοση και πολύ συχνά επίσης χρειάζεται και ένας χώρος. Τι διαπιστώνω, μόλις ε, στηθεί κάποιος ως ελεύθερος επαγγελματίας, και έχει ολοκληρώσει όλες τις διατυπώσεις. Ε, αυτό που ζητούν οι νέοι επιχειρηματίες είναι κάποια συνοδευτική βοήθεια. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και απόψη συμβουλών και ανταλλαγής απόψεων. Παρατηρούμε ότι για παράδειγμα στα φυτόρια έχουμε νέους δημιουργούς επιχειρήσεων με υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Δεύτερη διαπίστωση, στην Ευρώπη έχουμε επιχειρήσεις που κλείνουν, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, πολύ αριθμές. Είναι επίγον να δώσουμε προτεραιότητα στη δυνατότητα κατάρτισης για την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων. Θα μπορούσε αυτό να ενταχθεί σε ένα σύνολο εκπαίδευση στον τομέα του management που θα επιτρέπει την ε, εκκίνηση μιας δραστηριότητας ε, επιχειρηματικής. Πολλές φορές έχουμε και διευθυντές επιχειρήσεων επιτυχημένους που νομίζουν ότι μπορούν να ξαναξεκινήσουν μια δραστηριότητα αλλά δεν λειτουργεί πάντα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει σωστά σε συνεργασία, για παράδειγμα, με οργανισμούς νέων διευθυντών. Ο συνάδελφος Ρούμπι τα είπε αυτά οι διευθυντές μπορούν να εκπαιδευτούν και να συμμετέσχουν σε αυτή τη δραστηριότητα. Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ταμεία που κινητοποιούμε για ορισμένε δραστηριότητες, υπάρχουν περιπτώσεις επιτυχίας και στις περιφέρειες των πόλεων, στις πιο λαϊκές περιφέρειες, με νέους που γίνονται ε, διευθυντές επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, βγαίνοντας από τα σχολεία επαγγελματική κατάρτισης. Να μην στοχεύουμε λοιπόν την επιχειρηματικότητα μόνο στα ανώτερα πανεπιστημιακά διπλώματα. Θα πρέπει να το οικοδομήσουμε κατά κάποιο τρόπο σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Εγώ θέλω να προτείνω να τονίσουμε την διασυνοριακή διάσταση, διότι από εμπειρία διαπιστώνω ότι σε περιοχές διασυνοριακές όπου υπάρχει μεγαλύτερη αγορά εργασίας οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν πιο εύκολα στις γειτονικές χώρες. Αυτά έχω να πω αγαπητοί συνάδελφοι. Θα μπορούσε ενδεχομένως η Κομισιόν να επιλέξει κάποιες επιτυχημένες δράσεις οι οποίες θα δείξουν ότι στην Ευρώπη δεν αποτυγχάνουμε διαρκώς με τα προγράμματα που έχουμε ότι έχουμε περιπτώσεις επιτυχίας που σχετίζονται με την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών κονδυλίων που επιτρέπουν σε κάποιον να λάβει πίστοση από μια τράπεζα. Εγώ πιστεύω ειδικότερα ότι χρειαζόμαστε αυτή την ανάλυση ώστε όπως επιθυμεί ο συνάδελφος Ρούμπικ να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίος εγγεγραμμένος ο συνάδελφος Μπερτότ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Ρούμπεκ που άγγιξε αυτές τις διάφορες πτυχές που σχετίζονται με τις δυσκολίες της επιχειρηματικότητας. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω όπως συνήθως ότι η επιχειρηματικότητα των νέων επιλύεται με δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, εμπορικές δραστηριότητες και σπάνια απευθύνεται σε κατασκευαστικές παραγωγικές δραστηριότητες. Θεωρώ συνεπώς ότι η επαγγελματική κατάρτιση και η άμεση σύνδεση μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων αποτελεί την καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων εφόσον θέλουμε να επενδύσουμε στις παραγωγικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες. Μόνο εφόσον υπάρχει μία ε, σταθερή παραγωγική δραστηριότητα υπάρχει περιθώριο για υπηρεσίες, για εμπόριο, για όλες αυτές τις πολυάριθμες ε, δραστηριότητες. Ε, στην Ιταλία έχουμε τεράστιο αριθμό τέτοιων δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη σύνδεση μεταξύ παραγωγής που μοιραία οδηγούν σε πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Συνεπώ, αν μπορέσουμε να δώσουμε κατευθύνσει για καλύτερη σύνδεση μεταξύ πανεπιστημίων και επαγγελματικών χώρων και μεγάλων επιχειρήσεων που σχετίζονται στενά με τις παραγωγικέ δραστηριότητες και προτείνω να κατευθυνθούμε και προ δραστηριότητες ναι μεν ενημερωτικέ, αλλά και διαφόρων τύπων δραστηριότητε, όπω πώς να τα βγάλει κανεί πέρα με τη γραφειοκρατία, με τη φορολογία με τις επαφές ε, με τα πιστωτικά ιδρύματα για να προσφέρουμε υποστήριξη σε αυτούς τους νέους μικροεπιχειρηματίες οι οποίοι μπορεί να χάνονται λιγάκι μέσα σε αυτό τον κικαιώνα αυτού του κόσμου που δεν γνωρίζουν. Θα πρέπει λοιπόν οι κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν ε, να εστιαστούν προς δραστηριότητες παντός είδους βασικής κατάρτισης για το πώς μπορεί κανείς να τα βγάλει πέρα όταν ε, στείνεται ως μικροεπιχειρηματίας ε, στις υπηρεσίες ή στο εμπόριο και κάτι πιο σταθερό όσον αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, ομιλία. Το λόγο έχει τώρα η Κομισιόν. Παρακαλώ. Υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν που θα ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Good morning. Um, my name is... Λέγομαι Μάρκο Σεράβιτς, αναφέρομαι στα θέματα της επιχειρηματικότητας 2020. Συζητάμε τα θέματα εφαρμογής, παρακολουθούμε τη συνέχεια που δίδεται και κάνουμε τις δικές μας αξιολογήσεις. Όπως είπατε όμως και άλλες γενικές διευθύνσεις όπως η ΕΑΚ, η Connect, η Απασχόληση ασχολούνται και αυτές οι διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα ίδια θέματα για κάποια από τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν. Αναφερθήκατε στο Εράσμος αρκετοί από εσά. Θα συμφωνήσουμε ότι ο στόχος του να έχουμε 10.000 ανταλλαγές μέχρι το τέλος της επόμενης δημοσιονομικής περίοδου είναι σωστό και θα πρέπει να δούμε και από εκεί και πέρα δυνατότητες ποσοτικής αύξησης και όχι μόνο ποιοτικής βελτίωσης. Προς το παρόν ο αριθμός αυτό είναι περιορισμένος λόγω των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Πάντως προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα χρήματα το ταχύτερο δυνατόν. Περιμένοντας βέβαια να δούμε και τι θα γίνει στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Για το ΚΙΚ αναγνωρίζουμε το θέμα αυτό, ε, ε, αλλά ταυτόχρονα το θέμα αυτό είναι ευθύνη και αρμοδιότητα και των κρατών μελών και στηρίζουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών. Έχουν και τις δικές τους στρατηγικές απασχόλησεις οι χώρες μέλη και γι' αυτό ζητάμε από αυτές να μας πούνε με ποιο τρόπο πιστεύουν ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Για τα startups Έχουμε φτάσει σε κάτω από 7 ημέρες κατά μέσο όρο για να ξεκινήσει μια επιχείρηση στην Ευρώπη. Μιλάμε για ε, εταιρείε περιορισμένης ευθύνης. Αυτές παίρνουμε σαν υπόδειγμα. Αυτό ισχύει για να ιδρυθεί η εταιρεία. Φυσικά απαιτούνται άδειε από εκεί και πέρα για να ξεκινήσει οι δραστηριότητες η εταιρεία, η επιχείρηση. Και τώρα εμείς ξεκινήσαμε με μία μελέτη η οποία θα εξετάζει τις περιόδους αδειοδότησης, γιατί σε κάποιες χώρες μπορεί να ξεκινήσει κανείς την επιχείρηση σε μία μέρα, σε τρεις μέρες ή σε εφτά μέρες, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να λειτουργήσει κιόλα. Και όπως είπαμε, εμείς θέλουμε να υπάρχουν όλες οι άδειε διαθέσιμες μέσα σε ένα μήνα. Σε ένα περίπου χρόνο θα είμαστε σε θέση να αναφερθούμε σε πέντε πρότυπα εταιριών. Έχουμε πάρα πολλές χιλιάδες ε, τέτοιου είδους αδειοδοτήσεις, ε, δεν μπορούμε να ε, καλύψουμε τα πάντα, αλλά θα προσπαθήσουμε με βάση πέντε μοντέλα να δούμε πόσο δύσκολο είναι να πάρει κανείς τις άδειε στην Ευρώπη και να δούμε πού υπάρχουν οι σωστές πρακτικές. Ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο και για την υποστήριξή του πρέπει να μιλήσουμε για την πιο μεγάλη, αν θέλετε, το μεγαλύτερο σύνολο των πρακτικών τις οποίες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Θυμίζω ότι μόνο το 6% των πτωχεύσεων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη οφείλεται σε λόγους απάτης, ενώ το 94% είναι για αντικειμενικούς λόγους και για λόγους συγκυριακούς. Και γι' αυτό από τους ανθρώπους αυτούς προσπαθούμε να μάθουμε ορισμένα πράγματα και να τα εκμεταλλευτούμε. Σχετικά με αυτό που είπε η κυρία Τροτμάν, οι επιχειρηματίες χρειάζονται πράγματι περισσότερο από χρήματα, όχι μόνον χρήματα θέλουν να έχουν μια σχέση με υποστηρικτικές υπηρεσίες όχι μόνο στην αρχή της λειτουργίας αλλά τα πρώτα τρία με έξι χρόνια. Υπάρχουν χώρες στις οποίες υπάρχουν τέτοιου είδους διαδικασίες και η επιβιωσιμότητα, το ποσοστό βιωσιμότητας των επιχειρήσεων ξεπερνά το 50% τα πρώτα πέντε χρόνια. Είναι θετική η έκθεση λοιπόν και γι' αυτό Πιστεύουμε και εμείς ότι και η εκπαίδευση είναι βασική για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η βελτίωση του περιβάλλοντος φυσικά του οικονομικού είναι το βασικό, αλλά δεν είναι το μόνο. Κανένας δεν ιδρύει ε, μια επιχείρηση μόνο και μόνο γιατί η συγκυρία είναι ευνοϊκή. Το κάνει γιατί έχει τις ικανότητες, τις γνώσεις, τη βούληση. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε με το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ για τα συμπεράσματα. Κύριος Ρούμπιχ, παρακαλώ. Äh, σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά, πολλές ερωτήσεις ε, ακούσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, ανταπόκρισή σας. Θα ήθελα να δώσω μία μικρή διευκρίνηση σε ό,τι αφορά το ΚΙΚ. Το θέμα είναι να περάσουν όλα αυτά στα σχολεία όλα αυτά τα μηνύματα. Αυτό είναι η βάση του ΚΙΚ, αλλά αυτό που δεν έχουμε είναι τεχνολογίες με τις οποίες πρέπει να περάσουν όλα αυτά στα σχολεία. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτές να επικεντρωθούμε στην τεχνολογία το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διδασκαλία και την εκμάθηση στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε λοιπόν τι ε, τεχνολογίες έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές νέες ε, εφαρμογές, για παράδειγμα, μέσα στον iPad για την εκμάθηση. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας δάσκαλος πρέπει να είναι στο σχολείο και να μην μπορεί να χρησιμοποιεί μια τέτοια εφαρμογή. Ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει λοιπόν τέτοια νέα τεχνολογία για να διδάξει. Θα πρέπει λοιπόν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο να διαμορφωθεί η διδασκαλιακή εκμάθηση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, γνώση η τεχνολογία πότε θα πρέπει να διδαχτεί, σε ποια ηλικία καλύτερο στο σχολείο. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να δράσουμε σε όλες τις κοινωνικές, σε όλα τα κοινωνικό επίπεδα, ιδιαίτερα σε αυτά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ενεργεία. Πώς μπορούμε να πείσουμε τους νέους να συνεχίσουν και να ξαναδώσουν όθηση στην ε, εκμάθηση και στην εκπαίδευση. Αυτό ισχύει και για τους δασκάλους και αυτοί θα πρέπει να ενταχθούν στην όλη διαδικασία και όλα αυτά υποστηρίζουν το σύνολο που θέλουμε να πατήχουμε. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε τον συνάδελφο Ρομπίχ να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών 5η ε, 6 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι, Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης και δίνουμε αμέσως το λόγο στον συνάδελφο Κόβας για το ζήτημα που έχει, για το θέμα που έχει με τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών. Ευχαριστώ. η διευκόλυνση των μεταφορών της, ε, για τη βελτίωση των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χρήση βελτιώσεων. Έχω κάνει προτάσεις έτσι ώστε να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση όλων των μεταφορέων και γι' αυτό οι επιχειρήσεις μέσω των αρμοδίων εθνικών αρχών θα πρέπει να διασφαλίζουν και τις, τους, ε, την διευκόλυνση του τρόπου χορήγησης ε, του πιστοποιητικού καταγραφής και την εναρμόνιση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Δεν θα πρέπει να θα συχνά σε αδικαιολόγητες απορρίψεις. Θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα διαθέσιμα μέσα όπως και η ηλεκτρονική υπογραφή και το σύστημα καταγραφής θα πρέπει να είναι ασφαλές, ισχυρό και πλήρως λειτουργικό πριν τεθεί σε λειτουργία ο συγκεκριμένος κανονισμός. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης ένας μηχανισμός ανταλλαγής στοιχείων ανάμεσα στις εθνικές αρχές των κρατών μελών. Αυτό θα διευκολύνει την διαμεθοριακή ε, ε, μεταφορά. Θα πρέπει οι ρυθμίσεις να είναι συμβατές με τις ισχύουσες οδηγίες, τους ορισμούς και τα επίπεδα. Ιδιαίτερα αυτό το οποίο προτείνεται από την IAEA. E η μεταφορά ραδιανεργού υλικού απαιτεί φυσικά κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις στον τομέα της φόρτωσης και στον τομέα της αποθήκευσης. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από το εύρος της οδηγίας. Απαιτείται η συμβατότητα του συστήματος καταγραφής με την οδηγία 96-29 Ευρατών ε, που συμπληρώνεται από επιπλέον πέντε συγκεκριμένες ε, οδηγίες για την έκθεση σε ιατρικά υλικά, ενημέρωση, ε, μεταφορά μη ενεργού, ραδιενεργού υλικού κτλ. Αυτές οι οδηγίες προλαμβάνουν την έκθεση σε ιονίζουσες μορφές ακτινοβολίας από ιατρικές χρήσεις, και βοηθούν στην εναρμόνιση των ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ένας μεταφορέας ζητεί να εγγραφεί στον κατάλογο, το ιστορικό του θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στις εθνικές αρχές οι οποίες χορηγούν το πιστοποιητικό, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη δυνατότητα παρακολούθησης της εκτέλεξης των δραστηριοτήτων. Ε, οι μεταφορές βραδιενεργού υλικού με εναέρια και θαλάσσια μέσα δεν καλύπτονται γιατί υπάρχουν ρυθμίσεις προς αυτό. Δεν υπάρχει ανάγκη λοιπόν να αναφερθούμε στις θαλάσσιες μεταφορές και στις εναέριες μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξερευνήσει τις δυνατότητες ε, ε, τις οποίες παρέχουν τα πιο αποδοτικά συστήματα ελέγχου στις διάφορες χώρες. Αυτή θα ήταν η πιο αποτελεσματική λύση που μπορεί να εφαρμοστεί τάχιστα. Ε, οι αερομεταφορείς, σαν παράδειγμα, έχουν ένα πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα. Το νέο σύστημα, το οποίο εμείς καθορίζουμε, έχει σαν βασικό στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την διευκόλυνση των επιχειρήσεων μεταφορών. Παρ' όλα αυτά τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα παριθμός 1. θα πρέπει να γίνει και μία έκθεση για τις επιπτώσεις της εφαρμογής της έκθεσης της οδηγίας αυτής από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία διετία μετά τη θέση της σε ισχύ. Θα πρέπει να υπάρξει μικρή γραφειοκρατική επιβάρυνση και γι' αυτό σας ζητώ να υποστηρίξετε τις τροπολογίες αυτές και εγώ φυσικά θα λάβω υπόψη μου τις δικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Μαρινέσκου τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η ιδέα αυτή να υπάρχει ένα ενερμονισμένο σύστημα για τη μεταφορά ραδιοενεργού υλικού στην Ευρώπη είναι κάτι το θετικό και θα ήθελα να, να πω στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν όλε οι λεπτομέρειε. Αλλά θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη θα είναι παρόμοια. Όλοι θα βασιστούμε στα ίδια δεδομένα σε ό,τι αφορά θέματα εφαρμογής. Τι θα γίνει με τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών. Θα είναι και αυτά παρόμοια και ίδια σε όλα τα κρατη γιατί μπορεί μία συγκεκριμένη αίτηση να μην παρουσιάζει προβλήματα σε μία χώρα, αλλά να παρουσιάζει ε, προβλήματα σε κάποια άλλη. Πείτε μου λοιπόν, είναι όμοιοι και οι ορισμοί σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού. Και τέλος, θα ήθελα να μου πείτε και τι ισχύει σχετικά με τη νομική βάση. Το 2008 έγινε κάποια δουλειά σε ό,τι αφορά τα επικίνδυνα υλικά βάσει της συνθήκης. Τώρα εξετάζουμε την μεταφορά ραδιενεργών υλικών στα πλαίσια της ε, Euratom. Νομίζω ότι επί της βάσης αυτής βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μάλλον ε, διαβούλευσης και όχι συναπόφασης. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κ. Βιντάλ Κουάντρας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την καλή του έκθεση που στοχεύει στην δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής των μεταφορέων ραδιενεργού υλικού. Βασικός στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η μίαση του διοικητικού βάρους, διατηρώντας πάντα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας από τις ακτινοβολίες. Νομίζω ότι ο κύριος Κόβατς έχει βελτιώσει σημαντικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί επιμένει στην ανάγκη η οποία υπάρχει έτσι ώστε τα πρότυπα και τα κριτήρια τα οποία ισχύουν ε, για την ε, λειτουργία και την δημιουργία του καταλόγου να ταυτίζονται και πρέπει να εναρμονιστούν τα κριτήρια αυτά. Εφόσον είναι κοινά τα κριτήρια αν δεν είναι μάλλον κοινά τα κριτήρια δεν μιλάμε για ενιαία αγορά και για ε, εναρμόνιση των κριτηρίων. Η εξέταση των αιτήσεων για την επιτάχυνση της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Μητρώου ε, πρέπει να υπακούει ακριβώς στα ίδια κριτήρια. Από την άλλη βέβαια θα μπορούσε να υπάρξει η, πρόκληση για τους μεταφορείς να πηγαίνουν και να κάνουν τις αιτήσει τους στις χώρες τις οποίες οι απαιτήσει είναι λιγότερο θα έλεγα σημαντικές. στις διάφορες ρυθμίσεις τις οποίες διευκρινίζει ο εισηγητής για την ένταξη στο Μητρό των Μεταφορέων. Είναι θετικός όπως επίσης και η δυνατότητα επικοινωνίας με τα σημεία επαφής και τις αρμόδιες αρχές είναι οι καλύτερες δυνατές προτάσεις. Η βάση λοιπόν της έκθεσης αυτής είναι πάρα πολύ σωστή. Συνδυάζει την ασφάλεια και την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων αυτών με τη μείωση των γραφειοκρατικών και διοικητικών βαρών και για μια ακόμη φορά συγχαίρω τον κύριο Κόβατς. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Είμαι διευθυντή ε, τη μονάδα που ασχολείται με αυτό το φάκελο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοβαξία, για την έκθεσή σα και εκτιμάμε ιδιαίτερα τι συστάσει σα. Μια παρόμοια συζήτηση λαμβάνει χώρο στο Συμβούλιο. Εμεί στη δική μα πρόταση έχουμε αναγνωρίσει ότι πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση για την ραδιοπροστασία και αυτό τώρα θα αναπτυχθεί περισσότερο όπως πρέπει κινείται, όπως φαίνεται στην κατεύθυνση που προτείνετε εσείς ότι θα υπάρξουν κοινά κριτήρια ως βάση για τέτοια εγγραφή σε Μητρώα καθώς επίσης και ως βάση επανελέγχου της εγγραφής σε Μητρώα αργότερα, το οποίο ζητάτε και εσείς, σωστά. Όσον αφορά την ανάπτυξη λογισμικού, έχουμε προβλέψει να εμπλέξουμε τις ομάδες εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών που θα εξετάσουν όλα τα ζητήματα που θέτεται μαζί με την Κομισιόν ότι στο το ε, σύστημα να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι λειτουργικό, να είναι φιλικό προς τους χρήστες ε, και σταθερό. Όσον αφορά το αίτημά σας για την ίδια διοντολογία, κοιτάμε αυτή τη στιγμή την υπάρχουσα νομοθεσία και προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν είναι ίδιοι οι ορισμοί και κοιτάμε και τις απαιτήσει ασφαλείας του ε, IA τις οδηγίες όπου μπορούμε να αντλήσουμε αυτές τις γνώσεις, ειδικότερα όταν μιλάμε για κοινά κριτήρια και εναρμόνιση. Ζητάτε για ιστορικά δεδομένα, ναι, αυτά μπορούν να φυλαχθούν σε ένα τέτοιο λογισμικό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε συμφωνήσει όλοι και σκοπός είναι να διατηρηθεί η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφορών εθνικών αρχών. Συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα με τα όσο λέει ο κ. Βινταλ Κουάντρας ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει εγγραφή σε μητρό χώρας με χαμηλότερα πρότυπα. Συνεργαζόμαστε με τους εμπειρογνώμους του Συμβουλίου ώστε να καταλήξουμε ελπίζουμε σε κριτήρια τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες. Όσον αφορά την νομική βάση έγινε πράγματι και γι' αυτό μια συζήτηση εμείς και εκεί υπογραμμίσαμε, το ίδιο έκανε και η νομική μας υπηρεσία, το επιβεβαιώνει ότι αυτό που προτείνουμε εδώ συμπληρώνει τα βασικά πρότυπα ασφιλίας. Συμπληρώνει σημαίνει ότι υπό το καθεστώς του κεφαλαίου 3 της συνθήκης ε, Euratom θα αποτελέσει τη νομική βάση και οι συζητήσει στο Συμβούλιο πιστεύω καταλήγουν όλο και περισσότερο σε κοινή συνεννόηση από αυτού. Επιβεβαιώνω λοιπόν, επιδιώκουμε ενιαία εγγραφή σε μητροαπλοποιημένη απλοποιημένη διαδικασία, αλλά και διατήρηση και ενίσχυση του υψηλού επίπεδου ασφαλείας, διότι αν εφαρμόζουν όλα οι αρχές τα ίδια πρότυπα σε όλες τις χώρες, θα βελτιωθεί η ασφάλεια και θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Πιστεύω ότι θα προσφέρει όλο αυτό προς τη θεμενή Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Σιγητής για τα συμπεράσματα, κύριος Κόβετς. szólását, tehát úgy látszik, hogy ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και την Κομισιόν. Όπως βλέπω υπάρχει συμφωνία για αυτή την έκθεση μεταξύ μας, όλων μας. Αυτό που απομένει να κάνουμε λοιπόν είναι η κυρία Πρόεδρος να ανακοινώσει την προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλη επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο εισηγητή. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών θα είναι η 3η 4 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διαταξής του πρωινού. Σχετίζεται με το θέμα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βιντάλ Κουάντρας. Ευχαριστώ παιδί πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε. Λάβαμε 358 τροπολογίες με διαφορετικές τάσεις για το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτό είναι ο κοινό στόχος μας ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό συζητάμε την πρότασή της. Υπάρχουν αρκετά σημεία πάνω στα οποία έχει υπάρξει μεγάλη προσοχή από πλευρά συναδέλφων. Το πρώτο σημείο είναι η συμπερίληψη ήμι ε, των διαφόρων παραγόντων. Δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις επιστημονικές μέχρι τώρα έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε μια κατηγορία παραγόντων ε, στην ε, ρύθμιση την ομοθετική αλλαγές στις αγορές, στα συστήματα καταγραφής στις χώρες παραγωγής. Όλα αυτά είναι θέματα μη στατικά, είναι θέματα τα οποία εξελίσσονται σε μικρό χρονικό διάστημα και μπορεί να αλλάξουν δραματικά οι παράγοντες αυτοί. Συνεπώς οι παράμετροι αυτοί, οι παράμετροι αυτοί, οι παράγοντες αυτοί δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο θα έλεγα χρήσιμοι στην φάση αυτή παρά για τη διαμόρφωση ορισμένων προτύπων. Κάτι το οποίο σε αυτή τη φάση και αναφέρομαι στους παράγοντες και είναι σε αυτή τη φάση κάτι το όχι ιδιαίτερα σταθερό. Δεύτερον, είναι να δημιουργήσουμε έναν, δεύτερο επίπεδο στόχο για προχωρημένα βιοκαύσιμα. Εγώ βάζω το 2%, άλλοι προτείνουν το 2,5% και κάποιοι οι οποίοι προτείνουν και 3%. Πάντως γενικά η ιδέα του να υπάρξει μια ειδική κατηγορία για αυτού του είδους τα προχωρημένα βιοκαύσιμα είναι κάτι το οποίο ε, θα έλεγα προκαλεί μια κάποια συνένεση. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε ε, το διαφορετικό ποσοστό, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προς διαπραγμάτευση. Το τρίτο είναι το ανώτατο όριο, το ανώτατο όριο του 5% για συμβατικά βιοκαύσιμα. Αν εμείς καθορίσουμε έναν στόχο για τις δεύτερης γενιάς βιοκαύσιμα, τότε δεσμευτικό ε, ε, ποσοστό, τότε δεν είναι ε, ανάγκη να βάλουμε ένα επιπλέον όριο για τα υπόλοιπα καύσιμα, εφόσον έχουμε δεχθεί το 5%. Υπάρχει έτσι και αλλιώς ένα στόχος 10% για το 2020 και θα καθορίσουμε και αυτόν τον δεύτερο επίπεδο στόχο, δεύτερο επίπεδο στόχο για τα προχωρημένα βιοκαύσιμα, οπότε στην ουσία παραμένει ε, το υπόλοιπο. Ας μην το παρακάνουμε λοιπόν σε επίπεδο διακανονιστικό. Κύριος Τούρμες εκτός μικροφώνου. Το όριο είναι 7 ή 7,5% δεν είναι 5%. Κοιτάξτε, σε επίπεδο ενιολογικό, λέει ο Βινταλ Κουάντρατς, είναι ότι θα θέσουμε έναν στόχο δεσμευτικό για τα προχωρημένα βιοκαύσιμα. Αυτό έμεσα είναι και ένας τρόπος καθορισμού ενός ορίου επίσης και για τα καύσιμα τρίτης γενεάς. Κάποιοι από εσά έχουν επίσης προτείνει ένα ανώτατο όριο για τα καύσιμα τρίτης γενεάς, υψηλότερο όμως του 5%. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, νομίζω όμως ότι μπορούμε να το συζητήσουμε. Να φτάσουμε στο 6 ή στο 7%. Είμαι ε, ανοιχτός στην διαπραγμάτευση όπως γνωρίζετε όπως πάντα. Τώρα στις ε, πολλαπλές μετρήσεις. Δεν υπάρχει γύρω από τις πολλαπλές μετρήσεις ομοφωνία στην Επιτροπή. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει, να προκαλέσει μάλλον το αντίθετο από αυτό για το οποίο στοχεύαμε. Αυτή η πολλαπλή καταμέτρηση παραδέχεται αν θέλετε ότι δεν πετυχαίνουμε το στόχο του 10% οπότε κοροϊδευόμεθα και θα καλύψουμε το κενό με τα ορυκτά. Έτσι τουλάχιστον κατανοώ εγώ τη διαδικασία. Εξακολουθώ να πιστεύω πάντως ότι ο στόχος αυτός για τις δεύτερης γενεάς βιοκαύσιμα είναι ο καλύτερος τρόπος για την πρόθεσή τους. Το πέμπτο είναι η αηφορία και τα κριτήρια της αηφορίας. Είναι καλές οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί έτσι ώστε τα κριτήρια της αηφορίας να περιλαμβάνονται στη νέα οδηγία και να καταστούν αυστηρότερα λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα των ηθαγενών πληθυσμών, Δεν θα πρέπει να υπάρξει έλλειψη αηφορία στους τρόπους με τον οποίο υπάρχουν γίνονται βελτιώσεις της γης μετά από εκμετάλλευση και σίγουρα εκεί θα βρούμε μία κάποια συνεννόηση και κάποια όρια. Αλλά για τα απόβλητα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια κριτήρια, εφόσον βέβαια ο ορισμός για τα απόβλητα είναι ο σωστός. Θα πρέπει εδώ να αποφύγουμε τις απάτες. Και τέλος, σχετικά με την αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων, ξέρετε ότι αυτή η αρχή δεν είναι απόλυτη. Η οδηγία για τα απόβλητα εξαιρεί ορισμένες κατηγορίες και υλικά μη επικίνδυνα που προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή από δασοκομικές εκμεταλλεύσεις. Και υπενθυμίζουν ότι η απόκληση από την ιεράρχηση αυτή μπορεί να είναι απαραίτητη για ένα συγκεκριμένο απόβλητο όταν αυτό είναι απαραίτητο και καλύπτεται για περιβαλλοντικούς λόγους ή για τεχνολογικούς λόγους. Λοιπόν αυτή είναι η γενική εικόνα στην οποία έχουμε φτάσει μετά από όλες τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει. Είδατε ότι σε ορισμένα σημεία υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης, και αυτό θέλω να κάνω, να σας ευχαριστήσω βέβαια και για την προσπάθειά σας και για το ενδιαφέρον το οποίο δείξατε στη συγκεκριμένη οδηγία. Μια οδηγία η οποία διανοητικά, αν θέλετε, οικονομικά και πολιτικά παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον και είμαι πεπισμένος ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία και θα καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο με τη βοήθεια όλων σας. Ευχαριστώ τον Βινταλ Κουάντρας η κυρία Βαν Μπρέμπτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σιγητά, συνάδελφοι. Παίρνω το λόγο εξ ονόματος ε, της Μπέρτα Τόμψον, της συγγητριάς μας, η οποία δεν μπόρεσε να παραστεί εδώ. Δεν πρόκειται να σας παρουσιάσω τις δικές μου τροπολογίες, αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των θέσεων των δικών μου και της σκιώδους Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις, ε, την έκθεση, για, τις, ε, για την εργασία σας. 400 σχεδόν τροπολογίες, μεγάλος λοιπόν ο όγκος της εργασίας που είχατε να αντιμετωπίσετε και αυτό αποτυπώνει τις διαφορετικές θέσεις. Να απευθυνθώ και να μιλήσω στα, για τα βασικά θέματα, για το 5%, το κάπου του 5%. Ίσως είναι σημαντικό να το θυμόμαστε ότι όταν το 2008 καταρτήσαμε την οδηγία για τις ανανεώσιμες αποφασίσαμε ένα στόχο του 10% για το στόχο λοιπόν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι για τα βιοκαύσιμα, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και να θυμόμαστε ότι, ότι σε ό,τι αφορά και την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, σκοπός ήταν να περιοριστεί ο όγκος των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στις μεταφορές. Αυτός ήταν ο στόχος και ξέρουμε ότι ασφαλώς υπάρχουν μεγάλε μεγάλες διαφορές μεταξύ των βιοκαυσίμων οι διαφορές μεταξύ εκπομπών του άνθρακα, μεταξύ βιοεθανόλη, βιοδίζελ κτλ. Αυτό θα πρέπει να λεφθεί υπόψη και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι χαμηλέ οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα μέσω αλλαγών της χρήσης. Έγιναν λοιπόν κάποιε αλλαγέ σε ό,τι αφορά το 10% σε ό,τι αφορά το ΚΑΠ είναι σημαντικό, θεωρούμε, να διατηρηθεί το όριο του 10% αλλά και το όριο του 5% σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά και αντιλαμβάνομαι ασφαλώς ότι οι επενδυτές έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις σε αυτή τη γενιά. Ιδιαίτερα στη δική μου εκλογική περιφέρεια να σας πω ότι ε, έχουμε πάρα πολλούς επενδυτές στην δική μου περιοχή και ασφαλώς αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει να προστατευτούν. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν αλλάζουν διαρκώς οι πολιτικές μας. Θα πρέπει να τις προστατεύσουμε αυτές τις επενδύσεις. Εκ παραλίλου έχουν γίνει έρευνες οι, οποίοι, οι οποίες έχουν καταδείξει ότι οι επενδύσεις μιας γενιάς μπορούν να μεταφραστούν με χαμηλό κόστος σε κέρδη. Ε, δεν είναι λοιπόν ε, αντιφατικά αυτά τα θέματα. Μπορούν να συνδυαστούν. Μιλάμε λοιπόν για τα προηγμένα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Συμφωνούμε λοιπόν με τον πολλαπλασιαστικό παράγοντα. Συμφωνώ ότι αυτός ο υποστόχος θα μας βοηθήσει. Και γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που έχουν γίνει διάφορες ε, προτάσεις στις αποτρολογίες για το 3% υποστόχο. Αυτό είναι πολύ απλό και διαφανές για τους επενδυτές. Είναι σημαντικό ο επενδυτής να νιώθει ασφάλεια. Αναγνωρίζετε γενικά ότι τα πιο προηγμένα βιοκαύσιμα δεν έχουν πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά το iLook, σε ό,τι αφορά δηλαδή και τα υπολείμματα. Γι' αυτό λοιπόν τα προηγμένα βιοκάψιμα δεν έχουν ουσιαστικά μεγάλη επίδραση στην τιμή των τροφίμων. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα κατάλοιπα φυσικά θα πρέπει να τηρούν και την ε, ιεραρχία. Είμαι βέβαιη ότι όταν λάβουμε τις ε, Τροπολογίε τις συμβιβαστικέ, τα πράγματα θα πάνε καλά και φυσικά προσβλέπουμε σε μια περαιτέρω επικοδομητική συνεργασία με τον συγκεκριτή και τους κοιοδείς. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Ρόντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοβάς για το εξαιρετικό του έργο για την ομάδα Άλτε και υπάρχουν τρεις κύριοι στόχοι η μέσων και η βελτίωσή τους για την προηγμένα βιοκαύσιμα δεύτερον επενδύσεις στην βιομηχανία των βιοκαυσίμων που υπάρχουν ήδη έχουν δημιουργήσει ήδη 300.000 θέσει στην Ευρώπη εργασίας και πρέπει να προστατευθούν και τρίτον η ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει να βελτιωθεί. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Άλντα ε, συμφώνησε με τον εισηγητή του κ. Βιταλ για τα στοιχεία κλειδιά αυτού του σχεδίου έκθεσης συμπεριλαμβανομένων ως δεσμευτικού στόχου για τα προηγμένα ε, βιοκαύσιμα, τη διαγραφή του πολλαπλού υπολογισμού έως ότου βελτιωθεί η επιστημονική γνώση επί του θέματος. Τα στοιχεία των υπολείπων τροπολογιών του ΑΛΤΕ προτείνει 2% στόχο ο κύριος εισηγητής για τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Εμείς προτείνουμε 2,5% ώστε να έχουμε φιλόδοξους στόχους και να αξιοποιήσουμε τις πλήρες δυνατότητες των βιοκαυσιμών αυτών. Δεύτερον, για να γίνει ο δεσμευτικός στόχος για τα προηγούμενα βιοκαύσιμα πιο αποτελεσματικός προτείνουμε ανώτατο όριο των συμβατικών βιοκαυσίμων στο 7,5% χωρίς τέτοιο ανώτατο όριο ανησυχούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις για τα προηγούμενα βιοκαύσιμα Επιπλέον το ανώτατο όριο του 7,5% θα διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις στη βιομηχανία για τα συμβατικά βιοκαύσιμα θα προστατευτούν. Επιπλέον, η συμβολή των βιοπροϊόντων και των πρωτεϊνών από την παραγωγή συμβατικών βιοκαυσίμων ε, στην αγροτική παραγωγή της Ευρώπης θα πρέπει να αναγνωριστεί. Διαφορετικά θα χρειαστεί να εισάγουμε από άλλα μέρη του κόσμου. Τρίτον, σχετίστε στενά με το 7,5% αυτό το ανώτατο όριο. Προτείνουμε μια τροπολογία με στόχο ένα διαφορετικό ανώτατο όριο εντός των όριων του συνολικού ο ανώτου για τα συμβατικά βιοκαύσιμα. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει συνένεση ότι η συμβατική βιοεθανόλη κατά μέσο όρο έχει καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το συμβατικό βιοντίζελ. Η τροπολογία προτείνει συγκεκριμένου στόχους για τη βιοεθανόλη κοντά στο 2% του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των μεταφορών. Αυτά είχα να πω εγώ. αν υπομνώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τον κύριο Κουάντρας και τους υπόλοιπους χειώδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Τούρμες. Παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Νομίζω το πρώτο θέμα που θα πρέπει να λύσει η νομοθεσία είναι το γιατί έχουμε θέσει αυτό το θέμα επιτάπητος. Επειδή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό το τμήμα της οδηγίας για τις ανεώσιμες, καθώς και το γεγονός ότι στις διαπραγματεύσεις αναφέρθηκε ότι μόλις η ILUC καταλήξει σε μια βρία συμφωνία, ότι υπάρχει έμεση χρήση γεών. Στη φάση αυτή λοιπόν θα πρέπει να δράση ο νομοθέτης. Το είπε και ο Αλέχο. Μου έκανε έκπληξη. Λέτε και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την πρώτη γενιά. Μπορεί κανείς να επιλέξει να αγνοεί τα προβλήματα. Νομίζω όμως ότι για την χάραξη πολιτικής είναι τόσο πασίφανες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε κάποιες χώρες του τρίτου κόσμου, ότι υπάρχει πρόβλημα με τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Άρα, μιλώντας, το να λέμε απλά λοιπόν ότι δεν υπάρχει έμεσος αντίκτυπος, τι να πω, αυτό δεν νομίζω ότι καταδείχνει σοβαρή αντιμετώπιση. Όσο δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ μας για το ότι υπάρχει πρόβλημα με τα καύσιμα πρώτης γενιάς, είναι αδύνατον να βρούμε οποιαδήποτε λογική λύση. Ελπίζω, ελπίζω και προκαλώ όποιον βγαίνει και διατείνεται ότι δεν υπάρχει έμεσος αντίκτυπος, να απαρνείται όλη την επιστημονική έρευνα που έχει γίνει από διεθνείς οργανισμούς. Τι λέτε ότι είναι ανοησίες αυτά που βγαίνουν και ε, διακηρύττουν οι διεθνείς οργανισμοί. Αυτά είναι πράγματα επί των οποίων θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Άρα, άπαξ και συμφωνήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να συζητήσουμε με ποιο μέσο θα επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Και φυσικά υπάρχουν προβλήματα, όπως η αλλαγή του κλίματος ή ο έμεσος αντίκτυπος. Στη τελική ανάλυση, προκειμένου να υπάρχει καλή εκτίμηση του προβλήματος, ουσιαστικά βασιζόμαστε σε κάποια μοντέλα σε κάποιες προσπάθειες μοντελοποίησης. Αυτοί που λένε λοιπόν ότι το μοντέλο του ILOC δεν είναι σοβαρό, τι να πω, προσεγγίζουν αν θέλετε ιδεολογικά αυτούς που λένε ότι δεν είναι σοβαρό το μοντέλο και το κλίμα. Ο κύριος Έλμερ δεν μου κάνει εντύπωση που μιλάει, γιατί αυτός αρνείται ότι υπάρχει οποιοδήποτε θέμα με το κλίμα, γιατί ενώ το 99% των επιστημόνων υποστηρίζουν ότι υπάρχει αντίκτυπος στο κλίμα, αλλά αυτό είναι κατά του μοντέλου, την το μοντέλο του iLook μπορεί να είναι λιγότερο ε, όριμο σε σχέση με αυτό του κλίματος, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε τουλάχιστον ότι η Αμερικανική Ομοσπονδιακή ε, κυβέρνηση αποδέχεται το μοντέλο του ILO και την έμεση αλλαγή χρήση γη ως βάση για την πολιτική της. και η Καλιφόρνια και το... η κυβέρνηση της Καλιφόρνιας το αποδέχεται. Το μοντέλο της Καλιφόρνιας είναι καλό, θεωρώ. Γιατί αναφέρει ότι η επιστήμη διαρκώ εξελίσσεται και γι' αυτό στην Καλιφόρνια έχει συσταθεί ένα συμβουλευτικό επιστημονικό συμβούλιο που διαρκώ εξετάζει τι γίνεται με, το κάθε, με την κάθε σοδιά προκειμένου να προσαρμόζονται οι πράξεις της πλέον πρόσφατες επιστημονικές ε, εξελίξεις. Άρα θα πρέπει σε αυτό το σημείο να συμπληρώσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειαζόμαστε ένα συμβουλευτικό επιστημονικό συμβούλιο που θα μας βοηθάει να προσαρμοζόμαστε στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Χρειαζόμαστε λοιπόν το ILOC. Δύο λεπτά, δύο λεπτά δώστε μου, Πρόεδρε, να κλείσω. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε το ILOC. Ίσως ο Αλέχο και κάποιοι άλλοι να πιστεύουν στην αγορά. Πιστεύετε, στην αγορά. Πιστεύετε, ε? Γενικά. Γενικά, γενικώ πω, πιστεύετε ότι η αγορά πετυχαίνει καλά αποτελέσματα από μόνη τη. Η έλλειψη συνεκτικότητα που χαρακτηρίζει την προσέγγιση σας είναι η εξή. Μία τράπεζα δηλαδή ή οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Πιστεύετε ότι μετά το 2020 Μπορούμε να θέσουμε έναν υποστόχο για τα βιοκαύσιμα δεύτερη γενιάς, αλλά πιστεύετε πραγματικά ότι θα υπάρχει αξιοπιστία σε ό,τι αφορά το στόχο αυτό, αν ε, χωρίς κάποιο χρονικό όριο. Όσο δεν έχουμε εισαγάγει το iLook, δεν υπάρχει κάποιο μέσο για να προσμετράμε την καλύτερη απόδοση των βιοκαυσίμων ε, δεύτερης γενναίας. Και έχετε δίκιο, Γιάννης, που λέτε ότι έχει καλύτερη απόδοση η βιοεθανόλη, αλλά χωρίς το iLook δεν θα ε, σε καμία περίπτωση αυτή η πρόοδος όταν αγοράζουν ε, οι εταιρείε τα βιοκάψιμα αυτά. Χωρίς την άλλη λοιπόν δεν θα υπάρχει αγορά ουσιαστικά για τα καλύτερα βιοκάψιμα δεύτερη γενιά που θα έχουν καλύτερη απόδοση και για την καλύτερη βιοεθανόλη. Δεν θα υπάρχει τέτοια αγορά, πολύ απλά. Και θα εξαρτώμαστε τελικά αποκλειστικά από τις πολιτικές αποφάσεις. 1,5, 2, 2,5 Τελευταία παρατήρηση. Ένα όριο 7,5% όπως αναφέρατε. 2,5% είπατε για τα βιοκάψιμα δεύτερης γενιάς. Να έχετε υπόψη ότι ο ηλεκτρισμός προσπαθούμε να προωθήσουμε μέσω της οδηγίας και τον ηλεκτρισμό στα αυτοκίνητα, στα γιοταχή και γι' αυτό είναι επίσης χρήσιμο να υπάρχει ένας ε, πολλαπλασιαστής. Μπορεί να έχουμε το 1,5-2% για τον ηλεκτρισμό. Το 7,5% πολύ απλά είναι υπερβολικά υψηλό ποσοστό στην όλη λογική. Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Τσίτσεστερ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Φοβόμουν ότι ο κ. Τουρμές θα τα έλεγε όλα και αυτό θα με λυπούσε. Θα χρησιμοποιήσω όμως τα δικά του λόγια. Είπε ανοησίες. Nonsense στα αγγλικά. Εγώ θα τη χρησιμοποιήσω στα πλαίσια της αυταπάτης. Εγώ υποστηρίζω το ζήτημα του iLook όπως το, του όπως αναφέρει ο κύριος συζήτητες. Το θέμα είναι τι μοντέλο θα χρησιμοποιήσουμε και με τι παραμέτρους. Στο κομπιούτερ μιλάμε για Geigo, για είσοδο έξοδο σκουπιδιών και αυτή η μεθοδολογία τώρα όσον αφορά το Outlook αυτό το 10% στόχος για τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας ποιο κομμάτι αυτού θα γίνει θα, σε ποιο ποσοστό αυτού θα συμβάλλει η ιστιοπλοεία γιατί εγώ είμαι μεγάλος ε, φανατικός της ιστιοπλοείας μιλάμε, Κλοντ μιλάω τώρα, μην με διακόπτεις άκουσα όλα αυτά που είπες ε, και θα τελειώσω σε ένα λεπτό. Αυταπατώμαστε με τη μεθοδολογία και φυσικά η μεγαλύτερη αυταπάτη είναι αυτός ο πολλαπλός υπολογισμός. Λέμε πολλές φορές ότι κάποια πράγματα θα προσμετρώνται πολλές φορές για το ενεργειακό τους περιεχόμενο. Αν αυτό δεν είναι αυταπάτη, τότε τι είναι. Να πω ότι υποστηρίζω τον εισηγητή και θεωρώ αξιόπιστη την εκθέσή του και είμαι βέβαιος ότι με τις αμίμητες ικανότητες του θα καταφέρει να βρει ένα συμβιβασμό. Καλό Σαββατοκύριακο, Κλοντ. Έλμερ, Συνάλφος Έλμερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να απαντήσω στον κύριο Κλοντ Τέρμες. Εγώ δεν αρνούμε την κλιματική αλλαγή, δεν αρνούμε μάλλον το ότι έχουμε κλίμα, ούτε το ότι αλλάζει, αλλά πρέπει να συζητήσουμε το γιατί. Θαυμάζω το πόσο εμπιστοσύνη έχει ο Κλοντ στα μοντέλα, δεδομένου ότι όλα τα μοντέλα κλιματικής αλλαγής ε, προτείνουν οι υψηλότερες θερμοκρασίες σύμφωνα με τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα ενώ στο σχετικό οργανισμό του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις της θερμοκρασίας τα τελευταία χρόνια παρά τη σημαντική αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Τώρα ο κ. Τέρμας ε, λέει ότι ο εισηγητής ε, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν έμεσες επιπτώσεις αυτών των προτάσεων. Δεν είπε αυτό είπε ότι υπάρχουν έμεσες επιπτώσεις αλλά ότι η επιστήμη δεν γνωρίζει ακόμα απόλυτα πώς θα λάβει αυτές τις έμεσες επιπτώσεις ως βάση για νομοθεσία. Και αυτό μου φαίνεται πολύ λογικό ως θέση. Συγχαίρω τον κύριο εισηγητή που θεωρώ ότι έκανε την καλύτερη δυνατή δουλειά στο πλαίσιο των σημερινών συνθήκων και του τρόπου σκέψης του παρόντος θεσμού αλλά μοιράζομαι και τι ανησυχίε κάποιων προλαλήσαντων όσον αφορά τι επιπτώσεις για τι βιομηχανίε, για τι επενδύσει και το βαθμό κανονιστική αβεβαιότητας που δημιουργούμε. Ερχόμαστε και λέμε ορίστε ένα στόχο 10%. Τώρα αποφασίσαμε ότι τόσο θα είναι ο στόχο. Επενδύστε λοιπόν τι απαραίτητε βιομηχανικές υποδομέ για το 10% και μετά από μερικά χρόνια θα πούμε α, ίσω κάναμε λάθο, δεν θα λέμε ίσως 10%, θα λέμε 5 ή 7% ή κάτι άλλο ένα από τα κύρια προβλήματα των βιομηχανικών επενδύσεων και της απασχόλησης στην Ευρώπη σε εποχές που τόσο πολύ τα χρειαζόμαστε είναι η ρυθμιστική, η κανονιστική αβεβαιότητα στην βιομηχανία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, ανησυχούν για την κανονιστική αβεβαιότητα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλό και θα πρέπει να σταματήσουμε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Θα με ευχαριστήσει ιδιαίτερα. Και στην πυρηνική ενέργεια λένε το ίδιο, ότι ε, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι η κανονιστική αβεβαιότητα. Δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι θα κάνει μεγάλε επενδύσει η βιομηχανία σε τόσο κρίσιμου τομεί για το μέλλον τη οικονομία μα, εάν συνεχίσουμε να αλλάζουμε διαρκώ του κανόνε. Νωρίτερα, κυρία Πρόεδρε, έκανε μια παρατήρηση ότι ο Σύγκριτης έκανε ό,τι μπορούσε καλύτερο δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, της του τρέχοντος τρόπου ορθόδοξη σκέψη, αλλά αυτή τη στιγμή ίσω τα πράγματα αλλάζουν. Είχαμε μια συζήτηση στο κοινοβούλιο για τον backloading, όπου είναι η πρώτη φορά που είδα να βάζουν επιτέλου μπροστά την απασχόληση και την ανάπτυξη. Είχαμε συζήτηση με οργανισμού ε, εργοδοτών και βιομηχάνων που λένε κάτι να γίνει για τι τιμέ τη ενέργεια, Το Συμβούλιο επιμένει ότι στην ανταγωνιστικότητα, τι φθηνέ τιμέ και την ασφάλεια τη παροχής ε, αντί να έχουμε αυτή την αιμονή με, το, ε, με την πράσινη οικονομία. Αποσύραμε το φόρο για, τις, ε, για τα αεροσκάφη, καταπληκτικό πράγμα, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή αμφισβητεί τις επιχορηγήσεις της Γερμανίας προς τις μεγάλες βιομηχανίες που ήταν απαραίτητες ως αποτέλεσμα του πολύ ψηλού κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και εγώ έχω να προτείνω στους συναδέλφους το εξή. Θα πρέπει να θυμάστε ότι σε οκτώ μήνες, ένα χρόνο, θα δούμε ότι αυτός ο τρόπος σκέψης, αυτή η αιμονή με την πράσινη οικονομία που έχει αναλώσει αυτό εδώ το κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια, θα αρχίσει να απαλύνεται, να αμβλύνεται και είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει σημαντικά η στάση μας. Ευχαριστούμε. Συνάδελφος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν ε, τον εισηγητή. Είμαι η εισηγήτρια ε, της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου. Να σταθώ λίγο σε αυτά τα οποία είπε ο εκπρόσωπος των Πρασίνων σχετικά με τις έμεσες επιπτώσεις των βιοκαυσίμων και της ε, αντίστοιχης οδηγίας η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Έχουμε βέβαια για την μόλυνση, έχουμε βέβαια ε, και για άλλες κατηγορίες. Αλλά το περισσότερο που μπορούμε να δεχθούμε είναι οι ρυθμίσεις στα πλαίσια του iLook. Είναι περίπλοκο, πρέπει όμως να υπάρχει ένα πρότοπο για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε την αηφορία. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό από το 2021 θα πρέπει να υπάρξει ένα κριτήριο αηφορίας ήδη από τη φάση των επενδύσεων. Έχουμε πρόβλημα όμως και με το ποσοστό, το, το ΚΑΠ το λεγόμενο. Generación que parece ser que es el que se produce desde los alimentos y cuánto le tienes que dar a segunda. Pero es que desde de segunda generación Λοιπόν, σχετικά τώρα με τα βιοκαύσιμα της δεύτερης γενιάς, οι ίδιες οι επιχειρήσεις λέγουν ότι ε, παράγουν τέτοιου είδους βιοκαύσιμα, αλλά παρόλα αυτά απαιτείται ένας χρόνος για να φύγουν από την καλλιέργεια των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς και να περάσουν στη δεύτερη γενιά. και από τους πράσινους έχει τεθεί και μέσω μιας τροπολογίας το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας ε, ε, που είναι μια, ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αναλύσουμε πιο προσεκτικά. Ένα άλλο θέμα, όπως είπα, είναι το θέμα της αηφορίας. Αυτό θα πρέπει να επιβεβαιούται από τις ε, χώρες μέλη και θα πρέπει να δούμε αν θα συμπεριληφθεί ή όχι στα κριτήρια της συγκεκριμένης οδηγίας. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Χέλμερ, ε, η υπερβολική διακανονιστική, αν θέλετε, η σωρία διακανονιστικών ρυθμίσεων είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει κανένα. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε την προσπάθεια σε ένα περίπλοκο ε, θέμα καταθέσαμε 103 τροπολογίες και προσπαθούμε να καταλήξουμε στα καλύτερα κριτήρια για αυτού του είδους την παραγωγή. Ευχαριστώ. Τροτμάνη, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ανησυχίες που με οδήγησαν στο να καταθέσω ορισμένες τροπολογίες. Η αηφορία των επενδύσεων πρέπει να έχουμε μπροστά μας τις ανησυχίες για την αηφόρο ανάπτυξη και, για το, και στην Επιτροπή μας, την Ήτρε και σε σχέση με τις επενδύσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί αν δεν γίνει αυτό δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα ε, για επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε ότι για το NER 300 αν δώσουμε λανθασμένες απαντήσεις σε αυτόν τον παράγοντα iLook τότε χάνουμε τα προγράμματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα σε σχέση με τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς. Οι τιμές για την ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών είναι πάρα πολύ υψηλές. Οι βιομηχανοί λοιπόν ανησυχούν σε σχέση με τη χρήση της βιομάζας. Θα ήθελα να έχουν ένα διοικητικό και διακανονιστικό πλαίσιο αξιόπιστο και θέλουν επίσης να έχουν και συγκεκριμένες προβλέψεις σε σχέση με τις χρηματικές ανάγκες. Γιατί αν δεν υπάρχουν και τα δύο αυτά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα ανταποκριθεί. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συνεκτική πολιτική ε, ευνοϊκή για τις ε, ανανεώσιμες πηγές και για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Ευχαριστούμε και όλους τους συναδέλφους σας που συμμετείχαν, έδειξαν πολύ ενεργό ενδιαφέρον κατά πάρα πολλές τροπολογίε σε ένα θέμα πάρα πολύ περίπλοκο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο σήμερα, προκειμένου για να απευθυνθώ, να, προκειμένου να απευθυνθώ σε κάποια από τα θέματα τα οποία ακούσαμε. Τα πιο σημαντικά. Σε ό,τι αφορά την, το αδιάσυστο των στοιχείων του iLook. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξόδεψε πάρα πολύ χρόνο για να κατανοήσει σε τι βαθμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη στην τρέχουσα μορφή της ως βάση για την ομοθετική πρόταση για το θέμα αυτό. Είδατε λοιπόν την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρήσαμε ουσιαστικά ότι η επιστήμη, οι αριθμοί, τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τη μοντελοποίηση του iLook είναι αρκετά στενερά, αδιάσυστα για να αυξήσουν τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων, αλλά όχι αρκετά αδιάσυστα για να αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα για το ποια βιοκαύσιμα θα θεωρήσουμε βιώσιμα, ποια βιοκαύσιμα θα επιδοτήσουμε κρατικά και το καθεξής. Και αυτή είναι ουσιαστικά η βάση επί της οποίας βασίστηκε η πρότασή μας. Θα πρέπει να το κατανοήσετε αυτό για να κατανοήσετε γιατί προτείνουμε και ένα κάπα, ένα το όριο. Γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια αντικατάσταση των παραγόντων, των παραπλασιαστών του ILUC, επειδή δεν ήμασταν σίγουροι ότι το μοντέλο ILOC θα ήταν ο απόλυτος τρόπος, ο απόλυτα σωστά τρόπος για να προχωρήσουμε και επειδή ανησυχούσαμε και για τη νομική βεβαιότητα που θα συνεπάγονταν, γιατί θεωρούσαμε ότι τέτοιοι πολλαπλασιαστές θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν και θα μπορούσε να γίνει διαφορετική μοντελοποίηση, η οποία θα οδηγούσε σε διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία και νομική ανασφάλεια εν τέλει. Γιατί αν κάποια άλλα μοντέλα ενδεχομένως καταδείκνυαν ότι υπήρχε διαφορετικός αντίκτυπος για τα βιοκαύσιμα, ενδεχομένως να κρίνονταν διαφορετικά η βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων αυτών από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό ήταν πάρα πολύ ατυχές. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ο πιο σωστός τρόπος θα ήταν να πούμε ότι κοιτάξτε το πρόβλημα είναι τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς που βασίζονται σε καρπούς που ε, παράγουν τρόφιμα και θα πρέπει να σταματήσει η ενίσχυση σημερινή. Αυτό ήταν το ε, σκεπτικό πίσω από το ανώτατο όριο του 5% για τα βιοκαύσιμα. Όχι για το πόσα βιοκαύσιμα θα μπορούσαμε να παράγουμε και να καταναλώνουμε, αλλά για το πώς προωθούνται αυτά τα βιοκαύσιμα η παραγωγή των βιοκαυσίμων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ο πλέον σωστό τρόπο. Κατανοούμε ασφαλώ και παρακολουθούμε τη συζήτηση και εδώ στην Επιτροπή, σε άλλε επιτροπέ, στο Συμβούλιο. Υπάρχουν και άλλε ιδέε. Να κοιτάξουμε ενδεχομένω και το στόχο, το, το ενδεχόμενο υποστόχο. Αλλά δεν είμαστε πεπισμένοι ότι ένας υποστόχος χωρίς ΚΑΠ θα επαρκούσε για να περιοριστούν με τον τρόπο που θα έπρεπε να περιοριστούν οι εκπομπές iLook. Και επανερχόμενος στο αδιάστητο των επιστημονικών στοιχείων, αυτό που μας λένε τα επιστημονικά στοιχεία είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό είναι κάτι το οποίο το διατρανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα είναι πώς θα ορίσουμε ποσοτικά το εύρος του προβλήματος και να κάνουμε διάκριση μεταξύ των ε, διαφόρων ζητημάτων. Παρακολουθούμε το τι συμβαίνει, τι εκτιλήσεται. Διαβάσαμε τις ε, τροπολογίες σε ό,τι αφορά την νομική βεβαιότητα που αποτελεί το κλειδί εδώ, ασφαλώς και θα πρέπει να βρούμε το συντομότερο δυνατόν μια λύση και κατανοούμε και μάλλον εκτιμούμε την ταχύτητα ε, προόδου του φακέλου αυτού και πραγματικά σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπινταλ Κουάντρας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν μέρος στη συζήτηση. Άκουσα με προσοχή τις παρεμβάσεις όλων σας. Είπατε κάτι με το οποίο συμφωνώ απολύτως και είναι κάτι το οποίο ισχύει και στην εκλογική σας περιφέρεια. Η σημασία που υπάρχει στην προστασία των επενδύσεων που έχουν ήδη γίνει. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση εμείς να διαταράξουμε μία ολόκληρη σειρά επενδύσεων και μία ολόκληρη σειρά θέσεων απασχόλησης που αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Και για το βιοδίζελ και για, το, και για την βιοεθανόλη τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν πρέπει να εξελιχθούν και δεν σκοπεύω να κάνω κάτι το οποίο να δημιουργήσει προβλήματα. Νομίζω ότι η διευκρίνηση αυτή ήταν απαραίτητη. Και οι προτάσεις σας επίσης δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτό το οποίο εγώ αρχικά είχα συμπεριλάβει στην έκθεσή μου. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι έχουμε αρκετά περιθώρια για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Έχουμε δηλαδή μια πραγματική δυνατότητα να αναζητήσουμε μια σαφέστατη σύγκληση εδώ. Και εδώ ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα λεγόμενα συμπροϊόντα. Δηλαδή, και το λέω στην έκθεσή μου, η ειδική επεξεργασία για τη βιοεθανόλη είναι κάτι το πάρα πολύ ε, προφανές και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σαν προοπτική. Άκουσα επίσης με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον Κλοντ. Ο Κλοντ πράγματι είναι μια προσωπικότητα η οποία μας προσφέρει πάντα πάρα πολλά γιατί έχει πολύ πρωτότυπες απόψεις και πολλές φορές ιδιαίτερα πιστικές απόψεις. Εγώ, ο Κλοντ, δεν αρνούμε το φαινόμενο της ύπαρξης του Άιλουκ. Υπάρχει το Άιλουκ και πράγματι έμεσα Υπάρχουν ε, επιπτώσεις στη Βραζιλία, στην Ινδονησία, στην Ασία γενικότερα. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στα αυστηρά επιστημονικά στοιχεία βέβαια. Το πρόβλημα είναι όμως το πώς θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο, πώς μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε και τι συμπεράσματα βγάζουμε από το φαινόμενο αυτό. Αυτό υπάρχει, οι έμεσες αυτές επιδράσεις είναι σαφείς. ένα πρότυπο, ένα μοντέλο στη φυσική, στη χημεία, στην οικονομία είναι πάντα προσωρινό και αποδεικνύει την ικανότητα που έχουμε να προσμετρήσουμε με ακρίβεια τα φαινόμενα το μοντέλο, το πρότυπο ακριβώς δείχνει αν θέλει στην μετριοφροσύνη του επιστήμονα. Δεν μπορώ να κάνω την αξιολόγηση όπως ακριβώς θα ήθελα. Δεν μπορώ να κάνω να καρποφορήσει η εξίσωση την οποία έχω προβλέψει. Αλλά αυτό λειτουργεί σαν να συνέβαινε αυτό δηλαδή το πρότυπο, το μοντέλο. Αλλά η πληροφόρηση που μας δίνει το μοντέλο δεν είναι επαρκής, είναι ενδεικτική και θα πρέπει να εκλειφθεί όπως ακριβώς είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή σαν πρότυπο. Εάν αλλάξουν οι συγκυρίες με τις οποίες διαμορφώθηκε το μοντέλο, αν γνωρίσουμε καλύτερα τη λειτουργία του συγκεκριμένου φαινομένου, τότε πράγματι το πρότυπο θα πρέπει να ξεπεραστεί. Και γι' αυτό τα πρότυπα θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ επιφυλακτικότητα και με προσωρινό βλέμμα. Απαιτείται παράλληλα να υπάρχει μια νομική βεβαιότητα γύρω από τη χρήση των μοντέλων αυτών και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μοντέλων αυτών. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό και πάνω σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Συνεπώς προσπαθούμε να μετριάσουμε λοιπόν αυτά τα περιφερειακά φαινόμενα. Πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε πρώτος να δώσουμε κίνητρα και όχι να απαγορεύσουμε και να δεσμεύσουμε. Δεύτερον, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τις υπάρχουσες επενδύσεις αλλά και τις μελλοντικές επενδύσεις. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την νομική ασφάλεια γιατί αν πραγματικά βγάλουμε από τη μέση τα κάψιμα πρώτης ε, γενεάς τότε δεν θα υπάρξει προσπάθεια επένδυσης ε, ε, των πολλών δυνατοτήτων, των πολλών εκατομμυρίων, των πολλών θέσεων απασχόλησης και στα νέα γενεάς βιοκάψιμα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να μην κλείσουμε τις προοπτικές οι οποίες υπάρχουν να προχωρήσουμε θετικά, με ρεαλισμό και με νομική βεβαιότητα και έτσι θα πετύχουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν αυτά έχω στο νου μου. Νομίζω ότι στις τροπολογίες τις πολλές που καταθέσατε υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που θα συμπεριλάβω στι συμβιβαστικές και έτσι θα καταλήξουμε σε κάποιες σωστές ε, λύσεις ε, και να δούμε αν θα πρέπει λίγο όλοι να συμφωνούν ή θα πρέπει πολλοί να συμφωνούν λίγο. Ευχαριστώ Βινταλ Κουάντρας. Τέλειωσε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 20 Ιουνίου του 2013. Οι εργασίες της Επιτροπής μας θα συνεχιστούν σήμερα το απόγευμα στις 3.